Κύριε Πρωθυπουργέ της Ιταλικής Δημοκρατίας, σας ευχαριστούμε πολύ γιατί δεχτήκατε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μας εκθέσετε τη δική σας άποψη και όραμα για το μέλλον της Ευρώπης από πλευράς Ιταλικής Δημοκρατίας. Η Ιταλία είναι μία από τις ιδρυτικές χώρες και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί μπορούμε να προωθήσουμε αυτή τη συζήτηση για το μεγάλο αυτό ζήτημα που αφορά 500 εκατομμύρια κατοίκους. Υπάρχουν θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος για τους Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς θέλουμε να είμαστε η δημοκρατική καρδιά της Ευρώπης. Έχουμε εκλεγεί άμεσα από τους πολίτες και δώσαμε μεγάλη μάχη για την αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1,1 στο 1,3. Όσον αφορά τους ίδιους πόρους. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της μετανάστευσης. Είμαστε υπέρ περισσότερων επενδύσεων προς την Αφρική για να επιλύσουμε το ζήτημα από τη ρίζα του. Εγκρίναμε μία πρόταση που υπάρχει επιτάπητος σχετικά με αυτό το θέμα και θα θέλαμε και εμείς να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαδικασία ως πρωταγωνιστής έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες προς νότον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται ιδιαίτερα από το προσφυγικό. Ως προς το Brexit, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσεται υπέρ των ε, πολιτών και της προστασίας τους που ζουν στις Βρυξέλλες, ζητήσαμε μία ουσιαστική αύξηση πόρων, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαρθρώσεων να ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης και ως προς την εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν τον προσωρινό πρόεδρο της ε, Βενεζουέλας, τον κύριο Γκουαϊντό. Ένα άλλο θέμα που ε, εντάσσεται στο πρόγραμμα της ε, κυβέρνησής σας επίσης, αφορά ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να μετράει περισσότερο μέσα στα πλαίσια του νομοθετικού του έργου πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Σας δίνω το λόγο για να μας πείτε τη σκέψη της ε, Ιταλικής Δημοκρατίας για το μέλλον της Ευρώπης. Tanto vi potete registrare per il catch the eye con eh, il Presidente del Consiglio. Όσοι θέλετε μπορεί να ζητήσετε να καταχωρήσετε το όνομά σας για το catch the eye στο τέλος της παρέμβασης ε, του Ιταλού Πρωθυπουργού. Onorevole Presidente Tajani, onorevole... Κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι πραγματικά τιμή για μένα να απευθύνομαι σήμερα ενώπιόν σας και το λέω με ειλικρίνεια για να περιγράψω το μέλλον της Ευρώπης ε, σύμφωνα με τις θέσεις της Ιταλικής κυβερνήσεως. Η δέσμευση για το μέλλον της Ένωσης μας ξεκινά με μια πραγματικά συγκινητική αναφορά στον Αντώνιο Μεγαλίτσι, έναν Ιταλό που όριζε τον εαυτό του ως ερωτευμένο με την Ευρώπη, που ήταν θύμα των επιθέσεων πριν από δύο μήνες στο Στρασβούργο της τρομοκρατικής βαρβαρότητας. Σε έναν παγκοσμιωμένο κόσμο, όπου η οικονομία φαίνεται πως ε, πήρε τα πάνω της σε σχέση με, το, με τα δικαιώματα και όπου η οικονομία απομακρύνεται ε, από τις θέσεις των πολιτών μας. Πρέπει να θέσουμε ερωτήματα για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρμοδιότητές της, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κράτη, τα κράτη-μέλη, δηλαδή μόνα τους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύνθετες παγκόσμιες προκλήσεις. Το κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι, περνά μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα φαίνεται ότι έχασε την ικανότητα να προχωρά η, συγκυρία, ιστορική συγκυρία που είναι πολύ σύνθετη είναι, αποτελεί μια πρόκληση για όλους μας ε, από τα διάφορα θεσμικά επίπεδα να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα. Όπως έκαναν στο παρελθόν και άλλοι που μας προκάτοχοί μας και εμείς τώρα καλούμεθα να καταβάλουμε μια κοινή προσπάθεια με πλήρη επίγνωση των ευθυνών μας. Έχουμε την ευθύνη να θέσουμε εκ νέου σε κίνηση το ευρωπαϊκό εγχείρημα επιτρέποντάς του να αποκτήσει αξιοπιστία και συνοχή για να αυξήσει την βιωσιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά του. Οι προκλήσεις σήμερα είναι νέες, σύνθετες, απαιτούν όραμα και αν μου επιτρέπετε και μία δόση δημιουργικότητας. Προϋποθέτουν ωστόσο κατά βάση επίγνωση της αποστολής μας στον κόσμο. Τα μεγάλα αιτήματα που πρέπει, στα οποία πρέπει να δώσουμε απάντηση είναι ερωτήματα ουσίας. Ποια Ευρώπη θέλουμε. Ποια Ευρώπη χρειαζόμαστε. Πώς βλέπουμε εμάς στην Ευρώπη. Αυτά είναι ερωτήματα που έχουν συνδυσιακό χαρακτήρα και απαιτούν μεγάλη, μεγάλη αυτεπίγνωση. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει εκλεγεί απευθεία από τους Ευρωπαίους πολίτες και που είναι αυθεντικός θεματοφύλακας της Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε και πρέπει να είμαστε ένας λαός. Ο ευρωπαϊκός λαός σε μια διαδικασία ενοποίησης που μας δημιούργησε μια κοινότητα πεπρωμένου πέραν οποιασδήποτε νομικής, ε, ε, νομικής αναγνώρισης. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βίωσε σημαντικές στιγμές πρόοδου εδώ. Η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης χαράχθηκε από βαθιές διαιρέσεις, από συγκρούσεις, από αντιπαραθέσεις που διαμόρφωσαν έναν ε, ε, μια εθνική ταυτότητα, πλου, εθνικές ταυτότητες πλούσιες, ε, πολυ, πολυ, πολυγλωσσικές και που όμως λειτουργήσαν και θετικά νομικά και κοινωνικά. Ενσωματώσαμε στα οικονομικά μας συστήματα, τα εκπαιδευτικά μας ε, συστήματα, την, ε, την κοινωνική μας νομοθεσία, δίνοντας χώρο σε κυριαρχίες και πηγαίνοντας σταδιακά από το κράτος στην Ένωση. Επιτρέψαμε στα, στους πολίτες των κρατών μελών να κυκλοφορούν ελεύθερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν ενιαίο νομικό χώρο. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων πολύ περισσότερο και από την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των ε, κεφαλαίων ήταν μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Σκεφτείτε ακριβώς το βάρος του, του εθνικιστικού μίσους που είχε πλήξει τον, την Ευρωπαϊκή Ήπειρο το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα και που οδήγησε σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Οι Ευρωπαίοι, ιδίως οι νεότεροι, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν αυτή την θεμελιώδη ελευθερία κίνησης, χάρη στα οποία μπόρεσαν με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν να αποκτήσουν πλούτο ε, πολιτισμικό ε, και εμπειρίες υιοθετώντα και ε, αντλώντας από διάφορες εθνικές εμπειρίες και από την ικανότητα να συμμετάσχουν σε, μια κοινή, σε ένα κοινό συνέστημα. Η διαδικασία δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού λαού ε, τροφοδοτήθηκε και, και από τα νομικά εργαλεία καρπό μιας πολιτισμικής διαδικασίας κοινή υιοθέτηση της μιας νομικής ταυτότητας, της δημιουργίας ενός ίντεμ, ενός, ε, ευρωπαϊκού δήμου. Το έργο στο πλαίσιο αυτό του, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ήταν καθοριστικός και για την εθνική συνταγματική διαμόρφωση. Μέσω αυτών δημιουργήθηκε ένας ευρωπαϊκός νομικός χώρος όπου μπορούσε να αναγνωρίσει τον εαυτό του πολίτης και να αναζητήσει προστασία μέσω ενός πλήρου ολοκληρωμένου συστήματος προστασία σε πολλά επίπεδα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου που στηρίζεται σε μια κοινή παράδοση συνταγματικών ε, ταυτοτήτων. Το εξελιγμένο αυτό σύστημα δικαιοδοτικής προστασίας ε, που εντάσσεται πλέον ε, με ανεξίτηλο τρόπο στην κοινή νομική κληρονομιά της Ένωσης αποτελεί μια πολιτισμική κατάσταση που πρέπει να προστατεύσουμε ακριβώς λόγω των ενάρετων συνεπειών που επέτρεψαν να μπορέσει συλλογικά ο Ευρωπαίος πολίτης να έχει την επίγνωση της Ευρώπης τροφοδοτώντας την ε, κατανόησή του ότι μετέχει σε ένα κοινό έχειν μετέχει, ότι μετέχει σε έναν λαό που, που περιλαμβάνει τα ίδια γόνιμα στοιχεία πολιτισμού. Παρόλα αυτά δεν καταφέραμε να γίνουμε ακόμα και πλήρως ένας λαός. Δεν είχαμε το θάρρος να οικοδομήσουμε ένα ε, ολοκληρωμένο μοντέλο που πέραν της ρητορική θα ενθάρρυνε την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δήμου. Ιδίως μετά το 1989 έλειψε με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια μία ένα πραγματικά πολιτικό όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία προοπτική στο μακρύ χρόνο, με πρόβλεψη στο μέλλον. Γι' αυτό, χωρίς την οποία το όνειρο τελματώνει στην άμμο και χάνει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ιδρυτικών πατέρων της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έλλειμμα λόγω του ελλείμματος αυτού ορίμα, του οράματος των τελευταίων 30 ετών η Ευρώπη περι, περιορίστηκε στο στην οικονομική της διάσταση που οδήγησε σε μείωση της ε, ρυθμιστικής προσέγγισης σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς, περιορισμό της κοινωνικής υποστήριξης και του, του, του κράτους πρόνοιας που αύξησαν συνολικά τις ανισότητες πλούτου και ανισότητες ευκαιριών. Ιδίω με την άφηξη της οικονομικής κρίσης, η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση υποστήριξε πολιτικές λιτότητας με στόχο αποκλειστικά να περιορίσουν τα, τα κρατικά ε, τα κρατικά χρέη και να κρατήσουν το ποσοστό πληθωρισμού του κοινού νομίσματος όσο χαμηλότερα γίνεται. Εις βάρος μερικές φορές και της κατανάλωσης με καταστροφικές συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή πολιτική ενώπιον αυτής της ε, οικονομικής κρίσης ε, φοβήθηκε την και έχασε σταδιακά την επαφή με τον λαό, καθιστώντας ολοένα και μεγαλύτερη την απόσταση, όχι μόνο γεωγραφικά, μεταξύ Βρυξελών και των περιφερειών της Υπήρου μας. Σταδιακά η πολιτική έχασε την νομιμοποιητική και αντιπροσωπευτική της διάσταση. Εμφανίζεται στους πολίτες ολιγαρχική και απόμακρη, αδύναμη να καταλάβει τις πραγματικές ανάγκες της ε, κοινωνίας. Έγινε, όπως σωστά το είπε η πολιτιολόγος Άννα Γελόνκα, μία τελετουργική παράμετρος κάλυψης παγκοσμιοποιημένων δραστηριοτήτων που εν γέννη είναι ακατανόητες και μυστικές. Η δυνατότητα άρνησης, η άρνηση που δείχνει ο ευρωπαϊκός λαός της ελίτ ε, απευθύνεται σε εμά, μας θυμίζει ότι η πολιτική που υποδουλώνεται στην οικονομία χάνει τις αρμοδιότητές της, χάνει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στα αιτήματα. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή αποφασιστική για την ιστορία της Ευρώπης. Μας αναμένουν καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον μας. Ο ευρωπαϊκός λαός έχοντας ξαναεμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας και ζητά επιτέλους να τον ακούσουμε. Ζητά να υπάρξει μια αποφασιστική αλλαγή της μεθόδου και της προοπτικής. Είναι μια ευκαιρία, πολύτιμη θα έλεγα, να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, να επενδύσουμε στην μείωση της, απόκ, της απόστασης μεταξύ κυβερνώνων και κυβερνωμένων που τροφοδοτήθηκε από τη σιωπή, την αδιαφορία και την προσπάθεια ελαχιστοκυποίησης του μεγέθους για να μειώσουμε την, ε, τον κίνδυνο εσωτερικής έκρηξης του κόσμου που βιώνουμε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την σύγκρουση. Πρέπει να είμαστε όμως σε να την διακυβερνήσουμε αυτή. Δεν πρέπει να αποπεριοριστούμε σε έναν στήρο συντηρητισμό που αρμόζει σε μια πολιοκυμένη πόλη. Αντίθετα, πρέπει να εκφράσουμε με νέες μορφές δημοκρατίας την ικανότητά της να καινοτομήσει αναλαμβάνοντας, αναλαμβάνοντας και τον κίνδυνο να εγκαταλείψουμε κάποιες ε, παρελθούσες βεβαιότητες, κάποια μοντέλα ανάπτυξης ή σχέσεις δυνάμεων που δεν ανταποκρίνονται πλέον με την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να αφήνουμε κοινωνίες φτωχοποιημένες που εξαρτώνται από, αβέβαια, από ένα αβέβαιο μέλλον. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση και σε εξέγερση με απρόβλεπτες συνέπειες όπως βλέπουμε σε διάφορα φαινόμενα σε διάφορες χώρε της Ένωση. Ο ευρωπαϊσμός του 21ου αιώνα, κατά την άποψή μου, προποθέτει αναπόφευκτα να ξανασκεφθούμε ριζικά τις μορφές και τους θεσμούς που χαρακτήρισαν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενωπή τα τελευταία 30 χρόνια. Απαιτούν επιγόντω μία αυθεντική σύγκληση που για κάποιους οδηγούν στο να επανέλθουμε στο αρχικό, στην αρχική εικόνα του ευρωπαϊκού οράματος. Η Ευρώπη που φανταζόμαστε θα πρέπει να είναι μια Ευρώπη που επιτρέπει να προχωρήσουμε, όχι μόνο που να σταθεροποιούμε, να σταθεροποιεί, ή προς όφελος των πολιτών. Η προς των αλλάζει γρήγορα. Οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες είναι εξαιρετικά ε, ασαφείς κάποιες δυνάμεις που δεν μπορούν να, να καταφέρουν να δημιουργήσουν πραγματικούς πόλους διεθνούς ε, επιρροής αυξάνουν παρά τα αυτά την επίδρασή τους. Στο πλαίσιο αυτό κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να παίξει μόνο του έναν σημαντικό ρόλο. Εξού και η ευχή για μια ενωμένη Ευρώπη με θέση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτός είναι ένας δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε με συντονισμένο τρόπο, με μια φωνή. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να μιλήσει στον κόσμο. Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλόδοξη, συνεκτική, είναι αναγκαία κατά βάση για να βελτιώσουμε την ικανότητά της να συνομιλεί με τις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου ίσως είχα πει στην πρώτη παρέμβασή μου ε, στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό, στην συζήτηση με την Ουάσιγκτον για να διαφυλάξουμε το στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεών μας. Εδώ πρέπει να αναδείξουμε αυτά που μας ενώνουν, βασικές αξίες και όχι τυχόν διαφορές και ελλείψεις κατανόησης. Ταυτόχρονα, μια ισχυρή Ευρώπη είναι αναγκαία για να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε το διάλογο με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην παγκόσμια σκηνή. Η Ρωσία και η Κίνα είναι μέρη οποιασδήποτε λύση στις βασικές παγκόσμιες κρίσεις, ακόμα και στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κερδίσει αν αποποιηθεί της δυνατότητας να συνεχίσει το διάλογο με τη Ρωσία και την Κίνα ή να αποκτήσει ή να υποστηρίξει τις, απο, τις ε, απομονωτικές τους ε, προσεγγίσεις. Πώς θα γίνει όμως αυτή η ισχυρή Ευρώπη που όλοι θέλουμε. Πρέπει βέβαια να, να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες ε, που μας, παρέχει, που μας παράχει η ΠΕΣΚΟ, η διαθρωμένη μόνιμη συνεργασία, προς μία ευρωπαϊκή άμυνα που δεν είναι μόνο ε, που δεν δημιουργεί προβλήματα στη σχέση μας με, την, με τον ΝΑΤΟ αλλά αντίθετα είναι και ένα θετικό συμπλήρωμά του. Αυτό επιτρέπει και μεγαλύτερη ασφάλεια των, πολιτών, των πολιτών μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσει να έχει στενούς δεσμούς στην άμυνα και την ασφάλεια με το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά τον Brexit. Βασική προϋπόθεση για μια ισχυρή Ευρώπη στον κόσμο είναι να εξασφαλίσουμε κατά βάση την αλληλεγγύη και τη συνοχή μέσω της συλλογικής ε, συνεργασίας των κρατών μελών. Η μετανάστευση και η οικονομική διακυβέρνηση είναι βασικοί πυλώνες για να υποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την ε, αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Οι αρχές αυτές δεν πρέπει να οδηγήσουν σε διαιρέσεις τα κράτη-μέλη. Αντίθετα, τα κράτη-μέλη πρέπει να έρθουν κοντά στα μεγάλα αυτά ζητήματα που πρέπει να είναι κομμάτια της ε, ευρωπαϊκής αλληλεγγύης τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ακριβώς την αδυναμία της Ευρώπης να προτείνει να λειτουργούμε με τρόπο ίσο προς ίσο μεταξύ των πλευρών. Η, το θέμα της μετανάστευσης ήρθε αργά στην Ευρώπη και χάρη στην Ιταλία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις ε, μεταναστευτικές ζωές ως μία επίγουσα ανάγκη, αλλά πρέπει να αποκτήσει μια σταθερή θέση με αποτελεσματικό τρόπο. Και απευθύνομαι σε εσά με μια έκκληση που την επαναλαμβάνω σε κάθε σύνοδο κορυφής και σε κάθε άτυπη συνάντηση στην οποία μετέχω. Δεν πρέπει να, να καθυστερήσουμε περισσότερο την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου της 28 Ιουνίου πέρυσι. Χωρίς μια αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών δεν τηρείται καν η, η αρχή της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αντιμετωπίζει σωστά και με τη σωστή προτεραιότητα τις πρωτογενείς μετακινήσεις και ε, δεν θα οδηγήσουν ποτέ στο να αντιμετωπίσουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Ο Άλτο Μόρο έλεγε ότι κανείς δεν μπορεί να επιλέξει να είναι στην Ευρώπη ή να είναι στην ε, Μεσόγειο, γιατί όλη η Ευρώπη είναι στη Μεσόγειο. Η αρχή αυτή πρέπει πάντα να είναι μπροστά μας, όχι μόνο για να αντιμετωπίζουμε τη σωστή προοπτική του ζητήματος της μετανάστευσης. Πρέπει να είναι μπροστά μας και εκεί που διακυβεύεται η ίδια η ασφάλεια της Ευρώπης. Η υποστήριξη της ε, πολιτικής, των πολιτικών εξελίξεων στη Λιβύη ή ο ρόλος της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Η Ιταλία τάσεται υπέρ του ρόλου μας και της δράσης μας στη Μεσόγειο. Επισκέφθηκα την Αλγερία και την Τινησία και είχαμε και τη διάσκεψη του Παλέρμου το Νοέμβριο πέρσι. Σύντομα θα επισκεφθώ το Μαρόκο. Πρόκειται για μια συνεκτική στρατηγική της Ιταλίας για να συνδράμουμε και εμείς στη σταθερότητα και σταθεροποίηση της κατάστασης, να αντιμετωπίσουμε τις αλλεπάλληλες κρίσεις προς συμφέρον όχι μόνο της χώρας μας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Η Ευρώπη, πέρα από την Μεσόγειο, θα πρέπει να επενδύσει σε αυτή τη συνεργασία για την Αφρική και υπέρ της Αφρικής. Διαφορετικά, ε, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους επαναπατρισμούς που χρειάζονται μια συντονισμένη δράση της Ευρώπης αλλά και των κρατών μελών μεμονωμένα. Αυτό αφορά συγκεκριμένες απαντήσεις. Το μέλλον μας στην Αφρική πλαισιώνει αυτή την προσέγγιση. Και εγώ είμαι πεπισμένος Γι' αυτό. Γι' αυτό επισκέφθηκα τον Νίγηρα και το Τσάντ στα μέσα του Ιανουαρίου. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στα πλαίσια των αξιών μας να προβούμε σε μία νέα προσέγγιση υπέρ της Αφρικής, ένα νέο μοντέλο συνεργασίας ως ίση μεταξύ ίσων, αναλαμβάνοντας αμοιβαία ευθύνες. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αμέτωχοι στο γεγονός ότι ο πληθυσμός της Αφρικής, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες φτώχειας παρά τους φυσικούς πόρους που διαθέτουν αντιστοίχως. Ούτε μπορούμε να είμαστε αμέτωχοι στο γεγονός ότι η αφρικανική η οικονομία χάνεται σε μερικές χιλιάδες υπεράκτιες επιχειρήσεις που επενδύουν σε φορολογικούς παραδείσους. Χαίρομαι γιατί η προτεραιότητα συνεργασίας με την Αφρική έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ τον Ζαν Κλοντ που έδωσε αυτή τη νέα όθηση για το κοινό μας μέλλον αναγνωρίζοντας αυτή την προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ε, βέβαια και εγγραφή πιστώσεων καθώς και νέους τρόπους παρέμβασης. Η Ευρώπη θα πρέπει να ε, γράψει έναν απογραφικό κατάλογο βέλτιστων πρακτικών για να έχουμε μια ίση συνεργασία. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό μέσα στα πλαίσια και του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 21-27. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα μέσα και εργαλειοθήκες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ε, ροές, ιδιαίτερα στις ε, χώρες διαμετακόμισης. Και αυτό αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 6 δις ευρώ δόθηκαν στην Τουρκία για αυτό το σκοπό. Το Trust Fund υπέρ της Αφρικής έχει ένα κενό 550 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης έχει μεγάλη σημασία και η εσωτερική διαχείριση της μετανάστευσης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία των παρακτήων μας ή την προστασία με βάση την σύνοριοφυλακή. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πρώτη χώρα μετανάστευσης, αλλά και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά. Οι μεταναστευτικές ροές δεν φτάνουν από μόνες τους. Έχουν κάποια αιτία, γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά. Ο κανονισμός του Δουβλίνου του, που εγκρίθηκε το 2017, τον Νοέμβριο του 2017, δεν επιλύει από μόνος του το ζήτημα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνδράμουν με αλληλεγγύη και υποχρεωτικά. Γι' αυτό στις 28 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μίλησε για την αρχή της αλληλεγγύης και της ίσης κατανομής αρμοδιοτήτων, καθώς και το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν βλέπουμε τις καταχρήσεις, το τι γίνεται με τις ανθρώπινες ζωές, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το δίκτυο των διακινητών που αποτελούν μεγάλη μάστιγα για την ανθρωπότητα και βεβαίως απειλή για την ασφάλειά μας. Ας μην είμαστε διχασμένοι, ας μην είμαστε ούτε ε, λαϊκιστές, αλλά ούτε υπέρ και της απόλυτης αποκέντρωσης. Σας έχουμε μία κοινή Ευρώπη, μία Ευρώπη της ενότητας και της ασφάλειας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν δίχασμοι μεταξύ περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε και για την ΟΝΕ, την ολοκλήρωσή της, τη στιγμή που υπάρχουν εμπορικές και οικονομικές εντάσεις που κλειδονίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αφορά και τα εθνικά χρέη ως ποσοστιαία αναλογία του ΑΕΠ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία επανισορρόπηση και επιμερισμός ευθυνών για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει αυστηρή λιτότητα. Με βάση το δημοσιονομικό νόμο του 2019 από την Ιταλική κυβέρνηση πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στις σωστές ε, αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις χωρίς να αποτελέσουν συσήφιο έργο. Έχουμε προωθήσει τη σταθερότητα και σταθεροποίησή μας μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού εγχειρήματος και φυσικά η Ιταλική κυβέρνηση θα προωθήσει αυτή την πορεία. Παράλληλα, η προώθηση των δημοσίων επενδύσεων μέσα στα πλαίσια του ρυθμιστικού δικαιοδοτικού πλαισίου οδηγούν σε ένα σε μια δυναμικότητα της εθνικής μας ε, οικονομίας. Η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να φτάσει σε μια εξισορρόπηση ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και το σχέδιο Juncker, το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκή αναγνώριση της ανάγκης της δημόσιας παρέμβασης υπέρ των επενδύσεων. Τι σημαίνει να αντιμετωπίσουμε τη λιτότητα, όχι ότι δεν κατανοούμε την χρηματοοικονομική σταθερότητα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική σταθερότητα και την αηφόρο ανάπτυξη. Ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ αναφέρθηκε στην ελληνική κρίση και το γεγονός ότι η λιτότητα ίσας ήταν υπερβολική και παρακινδυνευμένη. Γνωρίζω ότι μερικοί σε ορισμένα χρόνια θα ζητήσουν συγνώμη επίσης για την έλλειψη αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ή της κοινωνικής Ευρώπης. Ήδη Σήμερα θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για την Ευρώπη του αύριο, ιδιαίτερα για τους νέους, για την εκπαίδευση, για τις καινοτομίες και για τις δημόσιες επενδύσεις που θα στρέφονται σε αυτούς τους στόχους. Γιατί μας ενδιαφέρει η αντιμετώπιση της, ε, του μεγαλύτερου ελλείμματος που υπάρχει. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική ενίσχυση και ανάπτυξη μετά από τη συνθήκη του Μάστριχτ και τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε να ε, διανύσουμε ακόμα πολύ δρόμο. Οι κρατικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει αυτή την πτυχή του ζητήματος. Το Eurogroup της 21ης Ιανουαρίου και η διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου όρισε μία ε, ομάδα υψηλών αξιωματών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και το θέμα των τραπεζικών κλειδονισμών και της Τραπεζικής Ένωσης. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις σε υψηλό επίπεδο. Και η εξηγίαση των τραπεζών είναι ύψης της σημασίας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν φτάσουμε σε μία νέα ύφεση πριν φτάσουμε σε μια νέα παλινοδία. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ ε, μιλάμε για την αντιμετώπιση των εθνικών χρεών, του εθνικού χρέους, σε σχέση 60% χρέος ΑΕΠ, χρέος ΑΕΠ. Αυτό είναι το όριο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η ΕΠΑ ΕΕ συνέδραμαν στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει να δημιουργηθούν κοινά μέσα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των κρίσεων συνδράμοντας με ευθύνη και αλληλεγγύη. Εάν δεν υπάρχει αρκετή αλληλεγγύη, μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί δεν έχουμε και μια κοινωνική Ευρώπη. Οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς αλληλεγγύης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα την ανεργία και την υποστήριξη της ανάπτυξης. Να δοθεί μια όθηση σε αυτές τις προτεραιότητες με, τη, με συγκεκριμένα μέσα και εργαλειοθήκες για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η διαφορά ανεργίας που πλήττει τους νέους που έχουν δυσθεώρητους δείκτες ανεργίας οδηγεί σε εθνικισμούς, σε εθνικιστικά στεγανά. Γιατί φυσικά οι χώρες που ευημερούν δεν θέλουν να αναλάβουν αυτό το κόστος, ενώ οι μειονεκτούσες περιφέρειες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια αηφορίας μία πιο δίκαιη και πιο ίση Ευρώπη θα πρέπει να αφορά και το επόμενο πι μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Να μην χάσουμε αυτή την προτεραιότητα. Με βάση και τις ε, υπαρξιακές μας προκλήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ των νέων προτεραιοτήτων μεταναστευτικό, ανάπτυξη, επενδύσεις, ασφάλεια και παραδοσιακές πολιτικές. Η ΚΑΠ θα πρέπει να τύχει της πλήρους υποστήριξής μας, καθώς και να προωθήσουμε την συνδρομή υπέρ μιας κοινωνικής Ευρώπης. Πολλές άλλες είναι οι προκλήσεις που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε να προωθήσουμε μια πιο, ένα πιο ίσο διεθνές εμπόριο υπέρ των καταναλωτών. Να προβάλλουμε κάθε πρωτοβουλία για να λάβουμε υπόψη και να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να συνδράμουμε στην προστασία των ηλικιωμένων και στην ψηφιακή εποχή, γιατί τα δικαιώματα ενέχουν και ένα κόστος. Η ε, Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένα security provider, λαμβάνοντας υπόψη και τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, έχει μεγάλη <coughs> σημασία το αρχικό μας μέλημα. Ποια Ευρώπη θέλουμε, ποια Ευρώπη χρειαζόμαστε, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, να μπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν μία ειρήνη που διαρκεί ήδη 60 χρόνια. Η απάντησή μου είναι για άλλη μια φορά η ίδια. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι κοντά στους λαούς της. Η Ευρώπη του 21ου αιώνα θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το σχέδιο υπέρ των λαών, με τους λαούς, για τους λαούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτό το συγκεκριμένο ρόλο ενίσχυσης του νομοθετικού έργου γιατί έχετε εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία, εκπροσωπείτε άμεσα τον Ευρωπαίο πολίτη και φυσικά υπάρχει και το θέμα λογοδοσίας έναντι των άλλων θεσμικών οργάνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές, αλλαγές ιστορικής σημασίας που άλλαξαν τα γεωπολιτικά δεδομένα. Παράλληλα, χρειάζεται μία ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας έτσι ώστε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων έναντι των πολιτών. Το ευρωπαϊκό σενάριο ορίζει ορίζει και ορίζεται από την απογοήτευση των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την στάση των πολιτών και αυτό αφορά και την Ιταλία που πολλές φορές δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς. Χρειάζεται αυτή η αλλαγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σωστή εκπροσώπηση θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αυτές τις αρχές. Σας δούμε το Brexit, θέμα ύψης της σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προσεχή χρόνια. Μπροστά σε αυτή την ε, πρόκληση η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενωμένη και αλληλέγγυα. Μετά από 60 χρόνια ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης χωρίς να υπάρχουν ε, χειροτικού τύπου αντιδράσεις. Πρόκειται για μία περίοδο χωρίς προηγούμενο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες και τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό που θα ανακύψει μετά από το Brexit. Κύριε Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να δούμε τι δεν λειτουργήσε σωστά και μέσα από τις συνθήκες και να αποφύγουμε τις φυγόκεντρες ε, δυνάμεις, όπως ισχύει και στη χώρα μου και είναι απότοκο της απογοήτευσης των πολιτών. Εάν θέλουμε η Ευρώπη να είναι το κοινό μας μέλλον, θα πρέπει να περάσουμε από το λόγο στην πράξη. Να ορίσουμε μια νέα Ευρώπη την Ευρώπη των λαών πιο αλληλέγγυα, πιο ίση, πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική. Τη μοναδική όπου οι πολίτες σήμερα και αύριο θα αξίσει να ζουν για αυτήν και μέσα από αυτήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Πριν δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κύριο Κατάινεν να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι για μας να μετέχουν τα κράτη-μέλη στις προσπάθειες ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση ζητούμε μια μεγαλύτερη δέσμευση στις επόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου ούτως ώστε να γίνουν δεκτές οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ενδεχόμενα κάποια, κάποιο συμβασμό για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Νομίζω ότι αυτά που λέω αντικατοπτρίζουν τις απόψεις όλων ε, στο, στο, στην Ολομέλεια. Ο κύριος Κατάινεν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, κύριε Πρωθυπουργέ Ταγιάννη, αξιότιμα μέλη. Η Ιταλία φυσικά ε, κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της Ευρώπης, έχει δώσει τόσο πολλά στην Ευρώπη. Είναι ιδρυτικό μέλος από την αρχή διαμόρφωσε την Ένωσή μας ε, σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Οι Σπινέλοι εν Ρώση είχαν ε, κρατούντο σε ένα νησί της Ιταλίας και εκεί εξεπώνησαν ένα σχέδιο για μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη. Κάλεσαν τα έθνη της Ευρώπης που τότε ήταν ε, αντιμέτωπα να συμμαχίσουν ούτως ώστε τα σφάλματα του παρελθόντος να μην επαναληφθούν. Μετά τον πόλεμο. Ο Ντεγκάσπερη έγινε ένας από τους ιδρυτικούς πατέρες της Ευρώπης. Και το 1957 στο Καπιτόλιο, στον λόφο του Καπιτολίου υπεγράφει η Συνθήκη της Ρώμης και δημιουργήθηκε η Ένωσή μας με έξι ιδρυτικά κράτη-μέλη. 60 χρόνια κατόπιν, το 2017, άλλη μια φορά, σε αυτά τα ίδια σκαλοπάτια της ε, Ρώμης, οι ηγέτες των κρατών μας στάθηκαν ο ένα δίπλα στον άλλον για να ανανεώσουν τη δέσμευσή του για την Ένωση. Αυτή τη φορά ήταν 27 από όλε τι γωνιέ τη Υπήρου μα. Αυτό είναι δείγμα του πόση πορεία έχουμε διανύσει. Το τονίζω αυτό γιατί η δική ιστορία της Ιταλίας είναι ένας από τους πολλούς λόγους που έχει μία τόσο μοναδική και σημαντική θέση στην Ένωσή μας. Αλλά επίσης γιατί καταδεικνύει ότι η Ευρώπη προοδεύει, ότι η Ευρώπη επιτυχάνει τα μεγαλύτερα επιτέγματα της όταν ε, έχει την Ιταλία και τους Ιταλούς ως παλόμενη καρδιά της. Η ιστορία αυτή πρέπει να μας βοηθήσει να είναι οδηγός και για το μέλλον. Για να υπάρξει ένα επιτυχές μέλλον για την Ένωσή μας, η ε, Ένωση χρειάζεται στην καρδιά της μια ισχυρή Ιταλία. Μια Ιταλία, από την άλλη μια χρειάζεται μια ισχυρή και πρωτοπόρα Ευρώπη. Πρέπει να οικοδομήσουμε από κοινού το κοινό μας μέλλον. Ενωμένη, και με αλληλεγγύη. Συνεργαζόμενοι πάντα και όχι αντιπαρατηθέμενοι. Συζητώντας και όχι ο καθένας για τον άλλον, σχολιάζοντας τον άλλον. Και αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματική ένωση αλληλεγγύης, η Ιταλία είναι το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσουμε. Εκεί ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για να βοηθήσει την Ιταλία να ε, ανοικοδομηθεί μετά τους τρομερούς σεισμούς του 1960. Κινητοποιήθηκαν πολλές χιλιάδες νέοι και εδόθησαν και 1,2 δισεκατομμύρια με βάση τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης. Όλοι είδαμε τις εικόνες αυτών των νέων εθελοντών από όλα τα μέρη της Ευρώπης που βοήθησαν να ξαναχτιστεί η αρχαία και επανέμορφη εκκλησία της Νόρσια. Αυτή είναι η αλληλεγγύη η οποία είναι η βάση της ε, ένωσής μας και πρέπει να συνεχίσει να είναι η βάση του κοινού μας εγχειρήματο. Η Ιταλία επέδειξε το ίδιο πνεύμα. Αμέτρητες φορές όλα αυτά τα χρόνια. Ο, πρόεδρο ο πρόεδρος Γιούνκερ το έχει πει επανειλημμένα. Η Ιταλία είναι ε, μία από τις χώρες που έσωσαν την τιμή της Ευρώπης ε, στην κορύφωση της ε, κρίσης ε, των προσφύγων. Γιατί ορισμένοι πόρισαν να στηρίξουν τις προσπάθειες της Ιταλίας. Αλλά επίσης είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη στο μεγαλύτερο μέρος της στήριξε όσο μπορούσε την Ιταλία. Από τότε που ξεκίνησε η μεταναστευτική κρίση μέχρι το τέλος του 2018 η Επιτροπή διέθεσε σχεδόν 950 εκατομμύρια για να στηρίξει τις ε, πολιτικές αυτές στην Ιταλία. 225 εκατομμύρια συγκεκριμένα δόθηκαν για επίγουσα βοήθεια για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης και να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις υποδοχής και να στηρίξει όλες τις αρχές και ε, τους πολίτες που βοηθούσαν. Η Ευρώπη στάθηκε στο πλευρό της Ιταλίας. Και να μην ξεχνάμε την επιχείρηση Σοφία ή το ρόλο της Ευρωπαϊκής Άκτο και Σύνορο Φυλακής που σώζει ζωές στη θάλασσα. Αυτό είναι μια κοινή προσπάθεια και γι' αυτό χρειαζόμαστε την Ιταλία. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να υπερβεί τις διαφορές της για να καταλήξει σε βιώσιμες και υπεύθυνε λύσεις. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να στηριζόμεθα σε ad hoc λύσεις. Βεβαίως έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που είχαμε την ε, κορύφωση, την κορύφωση της κρίσης όπου 80% ε, των ε, προσφύγων έφταναν ε, στην κεντρική Μεσόγειο. 7.000 ζωές σώθηκαν στη θάλασσα. Αλλά τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή, να κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές στο σύστημα ασύλου μας. Η Επιτροπή έχει υποβάλει πολλές προτάσεις και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να συμμετάσχει πλήρως η Ιταλία αν θέλουμε να επιτύχουμε σε αυτό το εγχείρημα. Αξιότιμα μέλη, κύριε Πρωθυπουργέ, Ευρώπη σημαίνει ειρήνη και ευημερία. Και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την υπεράσπιση των αξιών τη. Όλοι μαζί. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να επιτύχει η Ευρώπη. Και σημαίνει επίση ότι πρέπει να αποφασίσουμε πού θα γίνουν οι επενδύσει για να έχουμε τη μεγαλύτερη επίπτωση στην καθημερινότητα των Ιταλών και των άλλων Ευρωπαίων. Γι' αυτό, τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε έναν δίκαιο και ισορροπημένο προϋπολογισμό για το μέλλον, που είναι πιο αποτελεσματικό και εστιάζει περισσότερο στα θέματα που ενδιαφέρουν και θίγουν τους περισσότερους συμπολίτε μας. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τριπλασιασμό των πόρων για την μετανάστευση και την ασφάλεια. Σχεδόν τριπλασιασμό. Σχεδόν 33 δι Και πρότεινε έναν πιο αποτελεσματικό προπολογισμό για την εξωτερική δράση, για να φτιάξουμε συνεργασία με τις χώρες της γειτονία μας και ευρύτερα. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ιταλία, που είναι χώρα που έχει αναλάβει τόση ευθύνη για τα θέματα αυτά. Θα επενδύσουμε ούτω ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόμα, πιο παραγωγική. Και κλειδί για την Ιταλία θα είναι το 50% αύξηση στην χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία και τα 9 δις για την ε, ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία για να γίνει στην Ιταλία η ψηφιακή μετάβαση. Η επένδυση στο μέλλον σημαίνει επίσης να επενδύσουμε και στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή πρότεινε διπλασιασμό του προπολογισμού σε 30 δις για το πρόγραμμα Erasmus που είναι σύμβολο για την κινητικότητα της Ένωσης. Θέλουμε να αυξήσουμε τη στήριξη σε όλους τους τομείς και για την ανώτερη εκπαίδευση και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το 2017 πάνω από 65.000 ε, Ιταλοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα Έρασμος. Το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα οικοδομήσει περαιτέρω επί των επιτυχιών του ε, προγράμματος Juncker. Η Ιταλία είναι μία από τους ε, δικαιούχους που έλαβε τα περισσότερα ποσά, πάνω κάτω 58 δις, που βοήθησαν την Ιταλική οικονομία και πάνω από 2.015 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν χρηματοδοτήσεις. Το σχέδιο Juncker έχει αυξήσει κατά πολύ τις ιδιωτικές αλλά και τις δημόσιες επενδύσεις στην Ιταλία. Είναι θετικό σήμα, γιατί δεν πρέπει να ε, πληρώνει πολύ ο φορολογούμενο αν μπορούμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Έτσι σημειώνεται διαφορά παντού στην Ιταλία. 70 εκατομμύρια ευρώ βοηθάνε να ανακαινιστεί το νοσοκομείο του Τρεπίζο. 200 εκατομμύρια θα βοηθήσουν το Ιντερνετικό δίκτυο και θα δώσουν κατάρτιση ε, στη χρήση του ίντερνετ σε 4 εκατομμύρια. Και 500 εκατομμύρια θα βοηθήσουν γενικότερα, ούτω ώστε 7 εκατομμύρια στην Ιταλία να έχουν ευρυζωνική σύνδεση. 7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Και το πρόγραμμα InvestEU μπορεί να κάνει ακόμη πολύ περισσότερα. Συνολικά θέλει να αμοχλεύσει 650 δις επενδύσεων. Όλα αυτά μπορούν και θα σημειώσουν ουσιώδη διαφορά και πρόοδο στην Ιταλία, επιτόπου και παντού στην Ένωση. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν είναι δύσκολο να υπάρξει ανάπτυξη σε πολλές χώρες γιατί υπάρχουν ε, παγκόσμιες αβεβαιότητες αλλά και σε ορισμένες και λόγω εγχωρίων ε, αποφάσεων. Για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζεται εμπιστοσύνη και στα νοικοκυριά και στους επενδυτές η ε, εμπιστοσύνη είναι στο, σαν το οξυγόνο. Αντιλαμβάνεσαι ε, ότι υπάρχει μόνο όταν ε, δεν υπάρχει επαρκές και αν δεν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη δεν γίνονται οι αναγκαίες επενδύσεις. Η επένδυση στην Ιταλία είναι πιο αδύναμη από το μέσο όρο τη Ένωση για πολλά χρόνια. Και αυτό είναι διαθωτικό πρόβλημα και δημιουργεί λιγότερε θέσει απασχόληση για του Ιταλού. Παράλληλα, όπω επανειλημμένα λέω, η Ιταλία είναι μεταξύ των πιο δημιουργικών οικονομιών στον κόσμο. Το μέλλον της χώρας σας είναι στα χέρια σας. Να κάνετε αυτό που είναι αναγκαίο για να αποδεσμευτεί αυτή η δημιουργικότητα και να δώσετε ένα περήφανο μέλλον στους Ιταλούς. Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι βουλευτές, περάσαν δύο χρόνια από τότε που υποβάλαμε το, τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, που ξεκίνησε τη συζήτηση που διεξάγεται τώρα για το τι θέλουμε να επιτύχει η Ένωσή μας τα επόμενα χρόνια. Πέντε εναλλακτικέ λύσει έδιναν ε, πέντε διαφορετικέ πορείε από τον οποίο μπορούσαμε να ε, αποφασίσουμε. Αλλά ό,τι και να επιλέξουμε, ορισμένα θέματα είναι σταθερέ. Και ένα από αυτά είναι ο κεντρικό ρόλο τη Ιταλία στην περαιτέρω πορεία τη Ένωση. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Ιταλία. Και η Ιταλία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη. Δεν είναι έκπληξη, ούτε σύμπτωση που οι πρώτες γραμμές της Λευκής Βίβλου ήταν για τον Σπινέλη και τον Ρώση και το μανιφέστο τους. Οπότε, οδεύοντας προς το μέλλον, πρέπει να εμπνεώμεθα όλοι από τους προκατόχους μας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή, πιο ενωμένη ένωση για τις επόμενες γενναίες. Όπως έκανε και εκείνη για μας, ευχαριστώ πολύ. Τώρα προχωρούμε στις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Βέμπερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινήσατε από την προοπτική του λαού. Εγώ είμαι τη Βαβαρία. Πηγαίνω στις εκκλησίες, στην εκκλησία, στα, στο νοσοκομείο, στο δρόμο, μιλώ με τους ανθρώπους και διαπιστώνω τα ίδια προβλήματα που αναφέρονται. Κοινωνική δικαιοσύνη, προοπτικές για τους νέους. Για να απαντήσουμε πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι πέραν αυτών που μας είπατε. Για να απαντήσουμε στα οικονομικά προβλήματα η Ιταλία, πρέπει να πούμε ότι η Ιταλία έχει σήμερα, είναι η χώρα με το μικρότερο ρυθμό ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα για την Ιταλία. Είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για την... Ε, είστε χώρα της ομάδας των 7, μια, μια κινητήρια δύναμη στην Ευρώπη. Τι πρέπει να κάνουμε. Στο ΕΛΚ πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις. Και είδαμε ότι η κυβέρνηση στην Ιταλία δεν συμφωνεί ούτε καν για την ολοκλήρωση ενός ήδη εγκεκριμένου έργου μεταξύ Γαλλίας, ε, Γαλλίας Ιταλίας η κυβέρνησή σας για εβδομάδες ε, στο ξεκίνημά σας συζητούσε για το αν θέλετε ή όχι να είστε μέλη στην Ευρωζώνη. Πιστεύουμε ότι μόνο με μεταρρυθμίσεις μπορούμε να χτίσουμε το οικονομικό μέλος, μέλος της χώρας σας. Και αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και άλλες ε, χώρες που στην Κύπρο, στην Ισπανία, στην Ελλάδα είδαμε ότι αν θέλεις μπορείς να αλλάξεις την αγορά εργασία, το δικαστικό σύστημα, το φορολογικό σύστημα για να δώσεις θέσει εργασία. Και στη Γερμανία τη χώρα μου η ατζέντα 2010 του, του κ. Σρέντερ θεμελίωσε την μεταρρύθμιση. Μεταρρυθμίσεις λοιπόν για το μέλλον. Στην κυβέρνησή σας η κυβέρνηση δεν, δεν προσβλέπει στο μέλλον. Επίσης θεωρούμε ότι ένας σταθερός προπολογισμό είναι κρίσιμο για μια ισχυρή οικονομία, κάτι που δεν βλέπουμε στην Ιταλία. Αυξάνεται το χρέος, αυτό βλέπουμε. Αυτά συνοπτικά. Οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωση στην Ιταλία επιπλέον είναι πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη ανάπτυξης στην Ιταλία και είναι ευθύνη όχι της Ευρώπης αλλά της Ιταλικής κυβέρνησης. Εμείς σεβόμαστε απόλυτα το ότι είσαστε μια δημοκρατική κυβέρνηση με εντολή από τους ψηφοφόρους σας. Είναι ευκολότερο ίσως να κερδίσει εκλογές ως ένα κίνημα κατά τον ελίτ από το να μείνει στην κυβέρνηση ως ένα κίνημα κατά τον ελίτ. Κάποιοι γίνατε ή φτάσατε να γίνετε νέες ελίτ μετά στην Ιταλία. Να υπογραμμίσω ένα δεύτερο θέμα για το, μεταν, για το μεταναστευτικό, το ΕΛΚ πιστεύει ότι η Ιταλία αξίζει την αλληλεγγύη της Ευρώπης, κατανοεί την οργή των πολιτών της Ιταλίας. Για πολλά χρόνια η Ιταλία ήταν μόνη της και γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε ένα μηχανισμό αλληλεγγύη για την, αλληλεγγύης για την Ένωση, αλλά είναι πρόβλημα για μας να βλέπουμε ότι ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έρχεται εδώ και μας λέει ότι το όργανο στο οποίο μετέχει δεν ε, υλοποιεί τις υποσχέσεις του. Εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό. Για τις εξωτερικές σχέσεις, να σε ευχαριστήσω που υπογραμμίσατε την ευρωπαϊκή μας προσέγγιση ε, στην απάντησή μας για τη Ρωσία. Η Ιταλική κυβέρνηση περιμένουμε να συνενέσει στις κυρώσεις. Από την άλλη, τις τελευταίες μέρες είδαμε τις συζητήσεις για την Βενεζουέλα. Για το ΕΛΚ έχουμε εκεί έναν δικτάτορα ο οποίος έφτασε στην έγινε στην εξουσία με αντιδημοκρατικές εκλογές, με τη βοήθεια του στρατού που εμποδίζει ακόμα και τη μεταφορά φαρμάκων στη χώρα του. Και απ' την άλλη έχουμε ένα ελεύθερο εκλεγμένο κοινοβούλιο που ζητά απλά το δικαίωμα να γίνουν νέες πρόορε εκλογέ για τη θέση του Πρόεδρου. Σε μια επιστολή που έστειλε σήμερα προς τους Ιταλού πολίτε, ο κύριος Γκουαϊντό ρώτησε γιατί η Ιταλική κυβέρνηση δεν, υποστηρίζει, δεν υποστηρίζει τις δημοκρατικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα. Θα πρέπει να απαντήσετε σε, αυτό, σε αυτή την επιστολή αν πιστεύετε σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής κάποιες γενικότερες ε, σκέψεις. Ευχαριστώ για την δέσμευσή σας να αναζητήσετε κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις. Είπατε σήμερα ότι η Ιταλία γίνεται πιο παρούσα, πιο φωνάζει περισσότερο στην στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η δυνατή φωνή στην ευρωπαϊκή συζήτηση μπορεί να δείχνει εγωισμό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι βούληση συνένεσης, γιατί αν φωνάζουν όλοι, μόνο θόρυβος γίνεται. Είπατε επίσης για την ανάγκη να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ λαού και ευρωπαϊκών θεσμών. Είστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι όλοι εδώ, η Λέγκα, ε, τα πέντε αστέρια, το, ε, το Δημοκρατικό Κόμμα, Όλοι είμαστε εδώ, όλοι είμαστε ε, εκπρόσωποι των πολιτών, δεν είμαστε η ελίτ. Εδώ είμαστε εκπρόσωποι των λαών και εδώ πρέπει να αποφασίσουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες το λόγο έχει ο πρόεδρος Ούντο Μπούλμαν. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ είναι το σπίτι της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ένας χώρος δημόσιας συζήτησης και ειλικρίνειας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ειλικρινείς δηλώσεις και να σας ε, ενημερώσω για τις ανησυχίες μου. Ανησυχώ όταν ε, η κυβέρνηση μιας συντηρητικής χώρας και η κυβέρνηση της 7ης βιομηχανικής δύναμης στον κόσμο οδηγεί το Ιταλικό έθνος όλο και πιο πολύ σε οικονομική και πολιτική απομόνωση. Αυτό γίνεται σήμερα. Ενώ έχουμε ένα πλαίσιο, μια εξωτερική συγκυρία, όπου από τη μία δεν μπορούμε πλέον να βασιστούμε στην Ουάσιγκτον όπως το παρελθόν και αντιμετωπίζουμε και νέες απειλές από τη Ρωσία. Η οικονομία σας οδεύει προς την ύφεση και βλέπουμε ότι η βιομηχανική σας παραγωγή πέφτει. Σε αυτή την κατάσταση λυπάμαι ιδιαίτερα από την ε, ε, άνευ νοήματος κλιμάκωση των εντάσσεων μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Μα τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, σε τι χρησιμεύουν. Γιατί δημιουργείται συγκρούσεις κάτι τέτοιο, το ξέρετε, κανείς δεν κερδίζει από τέτοιες συγκρούσεις. είναι μια κατάσταση όπου όλοι θα χάσουν. Και η χώρα σα και η Ευρώπη. Ο πληθυσμό και των δύο χωρών μπορεί να πληρώσει υψηλή τιμή. Η Ιταλία και η Γαλλία είναι ο καθένα, ο δεύτερο εμπορικό εταίρο του άλλου. 17,6 δι είναι το ύψο του, ε, ε, ε, του ετησίου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Εκατοντάδε χιλιάδε θέσει εργασίας εξαρτώνται. Και αυτέ οι θέσει εργασία δεν είναι των ελίτ. Είναι απλών ανθρώπων και ο Ιταλικός λαός ε, δεν μπορεί να χάσει περισσότερο θέσει εργασία. Η Ιταλία φέτος θα αυξηθεί μόνο κατά 0,8%. 0,8% το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Μπορείτε να τα παρουσιάζετε αυτά ε, λέγοντας ότι θέλετε να επανέλθει η αξιοπρέπεια της εργασίας. Ε, δεν βλέπω όμω να οδεύεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν βλέπω να επανέρχεται η αξιοπρέπεια της εργασίας. 75.000 ε, εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους και πολύ περισσότεροι είναι σε επισφαλής και χαμηλόμιστες εργασίες ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταλείπουν τη χώρα σας ψάχνοντας για μια καλύτερη ζωή και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά οι οικονομίες των Ιταλικών οικογενειών τέθησαν εν κινδύνων με μία, λόγω μιας εσκεμμένης αντιπαράθεσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προπολογισμό σα. Ήταν αναγκαίο αυτό ή ήταν μόνο μία προσπάθεια προπαγάνδας ενό και μόνο ανθρώπου. Αυτό κόστισε στου Ιταλού 1,7 δί μόνο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών. Και γιατί, ούτω ώστε ο Σαλβίνη να έρχεται και να κάνει φιγούρα στι Βρυξέλλε. Ο οποίο έχει έναν αποδιοπημπαίο τράγο για όλου. Αλλά καμία λύση για τίποτα. Αυτή είναι σήμερα η Ιταλική πραγματικότητα. Από αυτό το οικονομικό χάος ο Σαλβίνη τώρα προσπαθεί να αξιοποιήσει την ε, μετανάστευση. Ήμουν πριν από δύο εβδομάδες στην Κατάνια και εκεί είδα ότι 47 άτομα, 47 άτομα για 12 μέρες δεν μπορούσαν να βγουν από το σκάφος που του είχε διασώσει. Το Sea-Watch. Μεταξύ αυτών ήταν και ανήλικοι και θύματα βασανιστήριων. Γιατί, γιατί, γιατί είχαν γίνει παιχνιδάκι μια κοινική πολιτικής. Αυτή δεν είναι η Ιταλία που ξέρουμε, συνάδελφοι. Γνωρίζουμε μια άλλη Ιταλία. Ξέρουμε τη μεγάλη ευρωπαϊκή Ιταλία του Αλτιέρο Σπινέλη, του Ντεγκάσπερη, που ποτέ, ποτέ για μικροπολιτικό υποτιθέμενο κέρδος δεν ε, ε έθεσαν εν κινδύνο την Ευρώπη ούτε τη χώρα τους. Καταλαβαίνω πολύ καλά και η ομάδα μου καταλαβαίνει πολύ καλά. Γιατί είναι απογοητευμένοι πολλοί πολίτες στην Ιταλία. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχε επιτύχει πολλά πράγματα είχε σώσει χιλιάδες και χιλιάδες από πνιγμό στη θάλασσα και η Ευρώπη δεν σας βοήθησε αρκετά. Δεν σας ε, επέδειξε επαρκή αλληλεγγύη. Αλλά ποιο σας απογοήτευσε. Όχι οι φιλοευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όχι εκείνοι που θέλουν να προωθηθεί η Ευρώπη. Κοιτάξτε, πείτε στους πολίτες σας ποιο δεν σας βοηθάει να κάνετε αυτέ τι μεταρρυθμίσεις. Είναι οι φίλοι του κυρίου Σαλβίνη. Είναι οι Κατσίνσκι και οι Όρμπαν και ο, ο Κούρτ στην Αυστρία. Αυτοί τα μπλοκάρουν όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πείτε την αλήθεια. Ενώ οι φιλοευρωπαίοι πάντα είναι στο πλευρό σας. Όταν ε, σώζετε ανθρώπους στη θάλασσα. Και είναι λογικό βέβαια αυτό να το κάνει. Υπάρχει ακόμη αυτή η Ευρώπη. Υπάρχει ακόμη αυτή η Ιταλία. Και οι δύο αγωνίζονται αυτή η θαυμάσια Ιταλία, αυτό το θαυμάσιο έθνος. Η Ιταλία του Σπινέλη και του Δεγκάσπερη. Αυτό βλέπω όταν βλέπω τους ψαράδες της Λαμπεντούζα που παρά τους νόμους Μπόση Φίνη ενώ ξέρανε τους περίμενε παρόλα αυτά συνέχισαν να σώζουν ανθρώπους στη θάλασσα. Το βλέπω στους ε, ε ναυτικούς του Ντετζότη που είναι ένα ε, σκάφος της Ιταλικής ακτοφυλακής που δεν έπρεπε να το κάνουν αλλά παρόλα αυτά είπαν ότι έχουμε έναν κώδικα δεντολογίας ε, των ναυτικών και το κάναμε και το βλέπουμε αυτά στους ε, δημάρχους που δίνουν κατάλημα και τροφή στους πρόσφυγες ακόμη και αν το αρνείται η κυβέρνηση αυτοί διασώζουν την αξιοπρέπεια της Ιταλίας αυτή είναι η τεράστια η θαυμάσια Ιταλία των ευρωπαϊκών αξιών αυτή την Ιταλία θαυμάζουμε σε αυτήν απλώνουμε το χέρι γιατί χρειαζόμαστε αλλά τότε θα πρέπει να σταματήσει η κυβέρνησή τους να φοράει αυτή τη μάσκα της απαθροπιάς. Γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική Ιταλία. Πρέπει επιπλέον να ξυπνήσει η, Ιταλία κατά τον η Ευρώπη κατά των λαϊκισμών, κατά αυτών που καταστρέφουν τις πατρίδες μας. Στην Ιταλία αξίζει η αλληλεγγύη μα. Η Ιταλία είναι στην καρδιά τη Ευρώπη. Μαζί με του στενότερους φίλου της. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Φίτο που θα μιλήσει από το ECR, θα ήθελα να πω στου ε, ε, εκπροσώπους πολιτικών ομάδων ότι αν υπερβαίνουν το χρόνο τους τον ε, μειώνουν από τους ομιλητές, από τους ανεξάρτητους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Και όπως ξέρετε πρόκειται για μια χώρα που έχει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Σε αυτό έχουν αναφερθεί πολύ. Ε, δεν έχει νόημα να κάνουμε μία γενική συζήτηση. Πολλές φορές οι διαγνώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την απτή πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να σταθώ στις επικρίσεις για το τι αποτελεί, από τι απαρτίζεται η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια σε, στον οικονομικό τομέα, στο μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό να δώσουμε ορισμένα στοιχεία σαφήνειας με συγκεκριμένα παραδείγματα, αντιφάσεις, τις οποίες θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Γιατί όταν μιλάμε για μετανάστευση, και τη στιγμή που η κυβέρνησή σας κατά αυτή τη θητεία προέβαλε μία δράση όχι τόσο αρνητική, αλλά ε, που προσπάθησε να βρει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους ε, ψαράδες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι όχι μόνο σώζουν ζωές, αλλά διαμαρτύρονται για θέματα που τους αφορούν εξαιτίας των πολιτικών μας. Ως προς το μεταναστευτικό, συμφωνούμε, αλλά τι θα γίνει με το σύμφωνο σταθερότητας. Εδώ υπάρχει μεγάλη ε, ανασφάλεια. Μιλήσατε στα Ηνωμένα Έθνη, ε, μιλήσατε για τη διάσκεψη του Μαρακές μετά στηρίσατε στάση αποχής για τη Βενεζουέλα. Μιλήσατε για ενιαία φωνή, αλλά στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ε, εξαιτίας της αρνητικής ψήφου της Ιταλίας δεν μίλησε η Ευρώπη με μία φωνή στα οικονομικά. Έχετε δίκιο ως προς την ανάλυση σας, αλλά τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματά σας είναι λανθασμένα. Δεν υπάρχουν επιλογές διαρθρωτικών πολιτικών. Αντίθετα, πολλοί λένε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος αύξησης του ελλείμματος εμείς το αυξάνουμε γιατί υπάρχουν πολιτικές που επιβαρύνουν τις δημόσιες δαπάνες. Μην μιλάμε ε, λοιπόν για διαρθρωτικές ε, αλλαγές. Σήμερα ζούμε δύσκολες στιγμές. Σήμερα μας μιλάτε για την ανάπτυξη και το ρόλο της Ιταλίας. Ο Υπουργός ε, Υποδομών σας θέλει να μας δείξει ότι το ΤΑΒ είναι ένα μεγάλο λάθος και θα πρέπει να μπλοκαριστεί. Πρόκειται για την γνωστή σιδηροδρομική γραμμή. Γι' αυτό θα πρέπει τα συμπεράσματά σας να οδηγήσουν στην πράξη. Και δυστυχώς η πράξη δεν οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση ούτε για την Ιταλία ούτε για την Ευρώπη. Από πλευράς φιλελευθέρων το λόγο έχει ο Γκί Φερχόφστατ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω Ιταλικά, Πρόεδρε. Γιατί πέραν της χώρας μου, μάλλον, κύριε Κόντε, είμαι ερωτευμένος με την Ιταλία και με τους Ιταλούς. Για μένα, η Ιταλία δεν είναι χώρα, είναι πολιτισμός. Είναι εκεί όπου γεννήθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και για αιώνες συγγραφείς, καλλιτέχνες, διανοούμενοι επισκέπτονταν την Ιταλία τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους για να ανακαλύψουν την Ιταλία το να ανακαλύψουν την Ιταλία σημαίνει να επισκεφθούν την Ιταλία να πάνε στη Φλωριντία, στη Ρώμη, στη Νάπολη ε, για να πεθάνουν. Ο Γκέτε αυτό έκανε και γι' αυτό κύριε Κόντε με πονάει κύριε Κόντε που βλέπω σήμερα την ε, πολιτική αποδυνάμωση της Ιταλίας κάτι που δεν ξεκίνησε πέρσι πριν από ένα χρόνια πριν από 20 θα έλεγα. Η εντύπωσή μου είναι ότι η πανέμορφη αυτή χώρασε πέρασε από το να είναι ένας από τους ιδρυτές της Ευρώπης και ένας από τους ε, υποστηρικτές της Ευρώπης στον τελευταίο τροχό. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω και εγώ και το Κοινοβούλιο και ο εξωκόσμος. Και αυτό δεν ξεκίνησε με τον Πρωθυπουργό Κόντε. Ξεκίνησε με την ε, κακή διακυβέρνηση της εποχής Μπερλουσκόνη και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το Μάλ αυτή η κακή διακυβέρνηση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας από τον Σαλβίνη, από τον Τιμάιο, τους πραγματικούς ηγέτες αυτής της κυβέρνησης μιας κυβέρνησης με συμπεριφορά μερικές φορές κύριε Κόντε αντιευρωπαϊκή και μερικές φορές με συμπεριφορά που έδειχνε μίσος κατά άλλων κρατών μελών, μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και η Ιταλική κυβέρνηση, η Ιταλική κυβέρνηση είναι αυτή που ε, εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί ενωμένη απέναντι στο Μαδούρο και να αναγνωρίσει τον Γκουαϊντό ως ε, προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας. Και το ξέρετε. Γιατί. Γιατί το κάνατε. Το κάνατε κάτω από την πίεση, του Κρεμλίνου, του Πούτιν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό μίλησε κάποιος γι' αυτό ήδη. Πρέπει να σταματήσουμε τον κανόνα ομοφωνία στο Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατό η Ιταλική κυβέρνηση δεν μετέχει στην πλειοψηφία του Συμβουλίου στην αλλαγή της ε, πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Ο κύριος Σαλβίνη θέλει να μπλοκάρει τα λιμάνια, ε, την είσοδο στα λιμάνια των μεταναστών, αλλά ταυτόχρονα μπλοκάρει την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Και για μένα αυτό είναι παράλογο, μια παράλογη συμπεριφορά, γιατί οι Ιταλοί πολίτες είναι οι πρώτοι που πληρώνουν την έλλειψη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτό. Αυτό είναι το τρίτο παράδειγμα που θα δώσω. Τον τελευταίο χρόνο εσείς, η κυβέρνησή σας, είστε υπεύθυνοι για την στασιμότητα και φοβάμαι αύριο την ύφεση της Ιταλικής και Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η κυβέρνησή σας έχει μόνο μία τακτική να ε, επανεκλεγεί κάνοντας δώρο χρέος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η τελευταία ελαφρότητα της κυβέρνησής σας, της κυβέρνησης από πλευράς Ντιμάιο που εκμεταλλεύεται τη θέση του για να υποστηρίξει τα ζηλέ ζών, τα κίτρινα γυλαίκα, ένα λαϊκιστικό ε, μοντέλο που υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που καίνε αυτοκίνητα, κλέβουν ε, μαγαζιά και καταστρέφουν στάσεις λεωφορείων. Ο Ντιμάιο συνάντησε το, τον Κριστόφ Σαλανσό. ο οποίος ζήτησε δύο φορές να γίνει πραξικόπημα κατά του εκλεγμένου Προέδρου της Γαλλικής ε, Δημοκρατίας. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Αυτό είναι μία ανεύθυνη συμπεριφορά. Όχι συμπεριφορά ενός αντιπροέδρου της κυβέρνησης μιας μεγάλης κοινοτικής χώρας. Πριν από ένα χρόνο, ίσως θυμάστε, στις 23 Νοεμβρίου του 2017, ο κύριος Ντιμάιο είχε στείλει μια ανοιχτή επιστολή στον Εμμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας το θαυμασμό του και πρότεινε το κίνημα, ότι το κίνημα των πέντε αστέρων ήταν ε, η, ιταλική εκδοχή του Αν Μάρς. Γελία συμπεριφορά. Η ερώτησή μου προς εσάς κύριε Πρωθυπουργέ είναι για πόσο καιρό θα είστε ο, ο χειράνθρωπος του Ντιμάιο και του Σαλβίνη. Σας καλώ σε κάτι εμπνευστείτε από τους λαμπρούς Ιταλικούς, Ιταλούς συμπατριώτες σας. Σπινέλη, Τσιάμπη, Ναπολιτάνο, Ντράγκη, ναι, ναι. Το Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, ναι. Ένα μεγάλο Ευρωπαίο με πραγματική ιδέα και μεγάλο άνθρωπο σε, αυτό το σώμα. Και μην ξεχάσετε τη φίλη μου Εμπαμπονίνο. Αυτοί είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που είναι το μεγαλείο της Ιταλίας και που έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κυρίου Κόντε και όλων αυτών των προσωπικότητων που ανέφερα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους ευρωβουλευτές ότι εδώ δεν είμαστε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ε, μιλάμε για τις ευρωπαϊκές προοπτικές και συζητάμε τις προτάσεις της Ιταλίας ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική. Το πολιτικό μου δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση Κόντε. Απλώς θέλω να έχουμε μία συζήτηση που να μην αφορά την κατάσταση στην Ιταλία. Γιατί δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησης. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά σας λέω ποιος είναι ο στόχος της συζήτησης. Λοιπόν, η κυρία Φορέντσα από την ΚΟΕ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ΚΟΕ θα ήθελα να υποβάλω ορισμένα ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας ως προς το τι θα συμβεί, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί στην Ιταλία. Δυστυχώς οι συνέπειες θα είναι πάντα ολέθριες, νεοφιλελεύθερες ε, πολιτικές ε, και ένα μεγάλο κύμα αντίδρασης και με τις δύο επιλογές φτάνουμε σε ολέθρια αποτελέσματα. Ε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους πληθυσμούς, τις γυναίκες, τους άνδρες, τη δυνατότητα δράσης, να καταπολεμήσουμε και να ε, ρίξουμε τα δεσμά του νέου φιλελευθερισμού. Να μιλάμε για ισότητα, γιατί μας πρόδωσε αυτή η κυβέρνηση Δυστυχώς ε, η σχέση ελίματος ΑΕΠ επιδεινώθηκε και ως προς το ίσο εμπόριο, ίσον όρον εμπόριο, δεν υπάρχει θέση της Ιταλικής κυβέρνησης για τη ΣΥΤΑ. Και νομίζω ότι η Ιταλική κυβέρνηση θέλει να φτάσει σε ε, ένα, ε, μια διαφορετική αντιμετώπιση των πλουσίων. Θα πρέπει να δώσετε μία απάντηση και για τη μεσημβρινή ε, Ιταλία. Επίσης, ως προς τον φυσικό αγωγό, τον διατλαντικό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μία ισότητα, να μην προσφέρουμε δωρεάν εργασία που πλήττουν την αξιοπρέπεια των Ιταλών. Η Oxfam μας δίνει απτά στοιχεία. Εσείς επιβάλλετε ένα flat tax, δηλαδή έναν καταποκοπή φόρο ανεξάρτητα από το εισόδημα. Μα αυτό είναι ο νέο και δεν μας απασχολεί μόνο αυτή η πτυχή του ζήτηματος. Στις 25 Οκτωβρίου 2018 μετά από ε, μία επίθεση της Casa Pound στο Μπάρι απαγορεύτηκε οι νεοναζιστές και νεοφασίστες να μπορούν να δρουν έτσι δημοσία. Πώς θα συνδράμετε στην εφαρμογή αυτού του διατάγματος και πώς βλέπετε τις σχέσεις του Υπουργού Εσωτερικών και των ε, εκπροσώπων της Casa Pound, που είναι ένα σχήμα νεοφασιστών και τίποτα άλλο. Η Χάνα Άρεντ μας το δίδαξε αυτό. Αυτή είναι η ρίζα της κακοδαιμονίας. Αυτός είναι ο φασισμός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Open Arms όταν διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπαμε ότι δεν μπορείτε να δράτε έτσι, θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Τα λιμάνια έκλεισαν για, τα, για τους 59 ανθρώπους που βρίσκονταν στην ανοιχτή θάλασσα. Τι κάνατε, τι κάνετε με την Τουρκία, δεν κάνατε τίποτα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου και υποχρεωτική relocation. Εσείς τι κάνετε. Επίσης, η ΜΚΟ δρούν στη θάλασσα. Εσείς στην ουσία τι κάνετε. Κρίνετε τις ΜΚΟ και τους αντιμετωπίζετε ως εγκληματίες. Δηλαδή στην ουσία εξισούνται η ΜΚΟ με τους διακινητές. Αυτό κάνετε. Η Άντα Κολάου, όπως και η Άντα Κολάου, θα ήθελα να σταματήσετε αυτή την ολέθρια πολιτική κλεισίματος των ε, λιμανιών και η δίωξη των ΜΚΟ. Τι μπορείτε να πείτε εσείς την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον της, αν ακολουθείτε μία τέτοια πολιτική κατά των ε, μεταναστών. Στις 8 Μαρτίου θα ε, δράσουν οι γυναίκες, οι φεμινίστριες θα κατεβούν στις πλατείες γιατί όταν αυτή η κυβέρνηση μιλά για τα δικαιώματα των ε, γυναικών κάνει το αντίθετο. Μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΦΑΜ βρέθηκε στην Ιταλία γιατί είδαμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να λάβουν το, χώρο, το λόγο οι γυναίκες. Τι γίνεται για τις ε, ε, γυναίκες, με τις γυναίκες της Ρώμης. Τι γίνεται με το Λουίτζι Σιέστα. Τι γίνεται με το σχέδιο κατά της βίας. Τι γίνεται με τον ελάχιστο ευρωπαϊκό μισθό. Έτσι θα μπορέσει να επαναξεκινήσει το μέλλον της Ευρώπης. Για να σώσουμε την Ευρώπη από το ναυάγιό της, θα πρέπει να έρθουμε αντίθετοι σε αυτές τις πολιτικές, αλλά και την πολιτική της κυβέρνησής σας. Σας παρακαλώ να μιλάτε πιο αργά, αν θέλετε να σας παρακολουθούμε, γιατί δυσχεραίνεται το έργο των διερμηνέων. γιατί στα Ιταλικά ειδικά πολλές φορές τρώμε τα λόγια μας, είναι δύσκολο για τους διερμηνείς. Τώρα ο Φιλίπ Λαμπέρ έχει το λόγο από τους Πρασίνους. Καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Στην Ιταλία, ε, η Ιταλία δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται καλά από το διεθνή τύπο, αλλά σκεφτόμαστε τη χώρα σας. Όταν σκεφτόμαστε τη χώρα σας έχουμε θετικές εικόνες στο μυαλό. Στην Ιταλία οι πολίτες ε, μαζικά ή εκφράστηκαν υπέρ του να μείνει η ίδρυψη δημόσια υπηρεσία. Στην Ιταλία εκφράστηκαν μαζικά υπέρ της ε, κατάργησης της ε, πυρηνικής ενέργειας. Στην Ιταλία δημιουργήθηκε το κίνημα για το slow food που είναι αντίδοτο στην ταχυφαγία που καταστρέφει, τα στομάχια μας και τις κοινωνίες μας. Και στην Ιταλία, χάρη στον ιστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργήθηκαν τρεις 3 εκατομμύρια πράσινων θέσεων εργασία. Όμω η κυβέρνησή σα, κύριε Κόντε, κάνει διαφορετικά πράγματα. Και μα θυμίζει τι χειρότερε στιγμέ που γνώρισε η πυρό μα ορισμένε φορέ. Όταν ο Υπουργό σα των Εσωτερικών, που μοιάζει να είναι ο πραγματικός, το πραγματικό αφεντικό, λέει ότι το όνειρό του είναι να απελαθούν οι Ρώμα από τη χώρα σα. Αυτοί που ζουν εκεί. Και επίση η χώρα σα θίγεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και μπορεί να αντιμετωπίσει και ύφεση. Και όπως ε, δείξατε και στην ομιλία σας, αποφεύγετε την ευκαιρία να κάνετε την οικολογική μετάβαση, την κινητήρια δύναμη της οικονομίας σας και την κινητήρια δύναμη της Ευρώπης. Θα μπορούσατε να επιλέξετε να ακούσετε τη, αυτούς που κρούν το κόδωνα του κινδύνου, όπως είναι η κυρία Μουρώνη, ή τους δημάρχους που είναι κατά των, κερδοσκοπιών, όπως η Ματήλ καζα Αλλά επειδή θέλετε να υπάρχει μια ξέφρενη ανάπτυξη, ξεκινάτε φαρανονικά και ανόητα προγράμματα όπως το τούνελ της ε, κοιλάδας του Χιούζ ή της, ε, περαιτέρου, του περαιτέρου τσιμεντόματος της χώρας από ορότερες της Ευρώπης. Αντιμετωπίζετε επίσης μια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Και εάν βεβαίως φέρουν και οι προκατοχοί σας ένα μεγάλο ποσοστό της ευθύνης, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το ότι η Ιταλία εφήγει από τις πολιτικές λιτότητες που υπάρχουν μετά τη συνθήκη του Μαστρίχτ. Αλλά αντί να επιδιώξετε να δημιουργήσετε συμμαχίες για να μεταρρυθμίσετε την Ευρωζώνη του ώστε το κοινό μας νόμισμα να ωφελεί όλα τα κράτη-μέλη, η κυβέρνησή σας τι επιλέγει. Αντιπαράθεση. Ε, δραματοποιεί την κατάσταση, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε τίποτα καλό και αυξάνει τους κινδύνους. Επίσης η χώρα σας είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του ασύλου και της μετανάστευσης. Θα μπορούσατε για την αξιοπρέπεια και την αποφασιστικότητα του Πιέρ του Μπάρτολο να είναι παράδειγμα. Είναι ο γιατρό στη Λαπεντούζα ή το ντομένικο Λουγκάνο που είναι ο δήμαρχος του Ριάτσο. Θα μπορούσατε να εμπνευστείτε από αυτούς. Αλλά δι' αυτό η κυβέρνησή σα θεωρεί ότι φταίνε οι μετανάστε για όλα τα δεινά τη Ιταλία και κλείνει την πόρτα στα καράβια που σώζουν την θεωρει οτι φταινε οι μεταναστε για ολα τα δυνάτια τη Ευρώπη, ε, σώζοντα Πρόσφυγε. Θα μπορούσατε να δράξετε το απλωμένο χέρι του Κοινοβουλίου που με πολύ ευρία πλειοψηφία ενέχνε την εγκατάλειψη των κανόνων του Δουβλίνου υπέρ τη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη που και εσεί και η κυβέρνησή σας ε, απαιτείτε. Διότι η μεταρρύθμιση που ενέχνε το Κοινοβουλίο μας ανταποκρίνεται ακριβώς στις απαιτήσει τη κυβέρνησή σα. Αλλά και εδώ το Τσίνκο Εστέλε αντιπαρατέθηκε εδώ κατά την ψηφοφορία. Ενώ η Λέγκα κρύφτηκε πίσω από την αποχή. Αντί γι' αυτό η κυβέρνησή σα προσπαθεί, αντί γι' αυτό, προτιμά αντί γι' αυτό, να συμμαχίσει με αυτού που είναι υπέρ του φρουρίου Ευρώπη, ενώ εγκαταλείπουν την Ευρώπη στην τύχη τη. Και ναι, μεν, το μεταναστευτικό είναι βέβαια θέμα για την Ιταλία. Είναι θέμα για την Ιταλία. Αλλά υπάρχουν δύο εκατομμύρια νέοι Ιταλοί, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεταναστεύσει ελεύθερα ή υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα του τα τελευταία 15 χρόνια. Πιστεύετε πραγματικά ότι οι αντιφατικές και συγκεκριμένες πολιτικές της κυβέρνησης θα τους ε, παρακινήσουν να επανέλθουν ή θα σταματήσουν την περαιτέρω διαρροή. Θεωρούμε ότι αν η Ιταλία γίνει κινητήρια δύναμη μιας ε, μετάβασης δημοκρατικής, ε, πράσινης και αλληλέγγυας θα δώσετε ένα μέλλον στη χώρα σας που είναι ανάλογο τη ιστορία τη, ανάλογο της θέσης που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά μας θα είμαστε εκείνοι που θα κινητοποιηθούμε γύρω από αυτές τις προτεραιότητες κάνοντας έκκληση ε, ε, επίγουσες ανάγκες για την Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας το λόγο έχει κυρία Ατζέα. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Κατάριν, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι η 17η συζήτηση που κάνουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Υπάρχει κίνδυνος να, ενώ όσο συζητούμε για το μέλλον της Ευρώπης να μην έχει παρόν η Ευρώπη. Εμείς συνεχίζουμε να θεωρούμε την Ευρώπη που ιδρύσαμε ως το σπίτι μας, αλλά η Ένωση χρειάζεται μια βαθιά μεταρρύθμιση, γιατί οικοδομήθηκε από την στέγη ξεχνώντας τα θεμέλια. Εμείς θέλουμε να δώσουμε στο σπίτι αυτό στέρεα και διαρκή και δυνατά θεμέλια. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο σωστή, πιο κοντά στους πολίτες, χωρίς να υπάρχουν κατηγορίες, χώρες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Θέλουμε να κερδίσει η πραγματική οικονομία την πρώτη θέση σε σχέση με τη χρηματοοικονομική προσέγγιση. Θέλουμε επενδύσεις, ε, ανάπτυξη, όχι λιτότητα. Θέλουμε μια Ευρώπη που να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και να μην υποκύπτει στις μεγάλες δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Κίνα και η ΕΠΑ. Θέλουμε μια ένωση όχι με όνομα αλλά στην πράξη. Και σα ρωτώ, αυτό σημαίνει να είμαστε υπέρ κατά της Ευρώπης. Πολλοί κοιτούν την ε, Ευρώπη, δεν ε, ε, βλέπουν το, την καμπούρα στην πράξη των άλλων, αλλά δεν βλέπουν τη δική τους πρώτα χτυπάνε την Ευρώπη και μετά αναγνωρίζουν ότι έκαναν μεγάλο, την Ελλάδα και μετά αναγνωρίζουν ότι έκαναν ένα μεγάλο λάθος. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να σημαίνει να αφήνουμε μια χώρα μόνο να διαχειρίζεται τη μετανάστευση. Το να είσαι ευρωπαϊστή σημαίνει να, δημι... να μετατρέψει φορολογικό παράδοσο... παράδεισο τη χώρα σου. Σημαίνει να αντιμετωπίζουμε σαν ε, πολεμική πράξη την εισαγωγή στην Ιταλία του, ε, ε, του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο που αφορά όλη την Ευρώπη. Αυτοί είναι ψεύδο-Ευρωπαίοι που έφτιαξαν μια Ευρώπη όχι των πολιτών αλλά των τραπεζών, τη γραφειοκρατίας και της λιτότητα μακριά από τους πολίτες. Μπορούμε να αλλάξουμε και πρέπει να μιμηθούμε την Ιταλία που αλλάζει αυτή τη στιγμή. Σε 7 μήνε καταργήσαμε τα, τις ισόβιες προσόδους των παλιών, ε, ε, βουλευτών, κόψαμε τις χρυσές συντάξεις, μειώσαμε τη φορολογία για τις μικρές επιχειρήσεις, ξεκινήσαμε να πληρώνουμε 30 δισεκατομμύρια χρέη των, του δημοσίου στους επιχειρηματίες. Σήμερα στην Ιταλία υπάρχει ε, ε, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Διαλύσαμε τη μεταρρύθμιση των συντάξεων που μας είχε επιβάλει η Ευρώπη για να έχουμε ε, σωστά νούμερα. Κύριε Κατάιν, εγώ είμαι από την Ούμπρια. Μιλήστε για την Ότσια. Στην Ότσια το μόνο που χρησιμοποιούνταν είναι να παίρνουν τα χρήματα των επενδύσεων για να τα μοιράζονται μεταξύ τους. Αυτό υποστήριξαμε στους πολίτες και αυτό κάναμε. Εμείς αυτό που λέμε το κάνουμε. Η πρόσφατη έκθεση για το 2019 για την Ιταλία που δημοσίευσε το Εουρίστες, γνωστό ίδρυμα, υπογραμμίζει την αύξηση της εμπιστοσύνης των Ιταλών προς την κυβέρνηση. 15 με 20 ε, ποσοστιαίες μονάδες πιο πάνω. Είμαστε μια κυβέρνηση αλλαγή, ακούμε τους πολίτες και τους παρέχουμε μια νέα ελπίδα για το μέλλον. Γι' αυτό μας κατηγορούν για λαϊκιστές. Κύριε Πρωθυπουργέ, όπως θυμήσατε. Αν αυτό σημαίνει να ακούμε τους, ε, να, να, αυτό σημαίνει να ακούμε τον κόσμο, ναι, είμαστε λαϊκιστές. Δυστυχώς πολύ συχνά σε αυτό το κτίριο, κτισμένοι στα, κλεισμένοι στα κλουβιά μας, ξεχνάμε να ακούμε τον, τους πολίτες. Ξεκινώντας από την κατάργηση της διπλής έδρας του Κοινοβουλίου, η δομή του, του χώρου στον οποίο είμαστε τώρα, που ερχόμαστε τέσσερις ε, μέρες το μήνα και κοστίζει 200 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε φίλοι των Γάλλων και δεν επιτρέπω σε οποιονδήποτε να μας δίνει μαθήματα για, την, για υποστήριξη σε ε, μπαχαλάκιδες. Εμείς δεν δεχόμαστε ότι μπορεί αυτό να θεωρείται αρνητικό. Εμείς δεν λέμε όχι στη δημοκρατία επειδή λέμε όχι στις δύο έδρες. Δεν, δεν σημαίνει όχι στη δημοκρατία γιατί είμαστε κατά ε, των δαπανών που κάνει το Κοινοβούλιο. Θέλουμε να μειωθούν οι τεράστιοι μισθοί των επιτρόπων που είναι πραγματικά κόλαφος για τους πολίτες. Για τις προνομιακές ε, συντάξεις των ευρωβουλευτών έχουμε ήδη υποβάλει μια πρωτοβουλία. Κύριε Ταγιάννη, υποστηρίξτε την πρότασή μας. Όλα αυτά δεν έγιναν μέχρι τώρα. Θα τα κάνουμε εμείς όμως χάρη στην ψήφο των πολιτών στις επόμενες ευρωεκλογέ και με την συνεργασία των άλλων δυνάμεων της αλλαγής. Έχουμε βάλει στην, στο τιμόνι της Ιταλίας μια πολύ καλή ομάδα τιμονιέριδων. Αυτό θα κάνουμε και στην Ευρώπη σε λίγο καιρό αλλάζουμε την Ιταλία, θα αλλάξουμε την Ευρώπη. Λοιπόν, προς γενική σας πληροφόρηση, θα ήθελα να σας πω ότι η επιλογή της έδρας δεν είναι αρμοδιότητας αυτού του σώματος ή των κρατών μελών που προσυπέγραψαν μια συνθήκη. Λοιπόν, κυρία Ατζέα, θα ήθελα να σας πω ότι εγώ δεν δέχτηκα τις 500.000 που μου προτάθηκαν στα πλαίσια της συνταξιοδότησης και δίνω αυτά τα χρήματα σε μία ομάδα αποτοξίνωσης ναρκωμανών. Η κυρία Πιτζότο, σήμερα κύριε Κόντε μας μιλάτε για την πρώτη πραγματική κυβέρνηση αλλαγών της Ευρώπης που με υπερηφάνεια μιλά για την εθνική μας κυριαρχία. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Έχουμε ε, το θάρρος να πούμε όχι στις Βρυξέλλες και στα προστάγματα του Βερολίνου. Δεν είμαστε υπέρ του μικρού Ναπολέοντα Μακρόν. Μια κυβέρνηση που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Ιταλών. Αυτούς τους μήνες η κυβέρνηση Λέγκα Πέντε Αστεριών έδειξε ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Ο Ματέο, ε, ο Ματέο Σαλβίνη μπόρεσε να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση και αντιμετωπίζουμε και την παράνομη μετανάστευση με την λεγόμενη κότα τσέντο προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το συνταξιοδατικό. Πολλά έχουν γίνει κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Να αυτονομηθεί το Βένετο, η Λομβαρδία, η Εμίλια Ρωμάνια, να γίνει μία μεγάλη φορολογική αναθεώρηση, να περικοπούν οι φόροι. Ο Μαδούρο είναι ένας μεγάλος δικτάτορας και είμαστε υπέρ με το λαό της Βενεζουέλας, Βενεζουέλας που θέλει την ελευθερία. Εμείς ε, ήδη εργαζόμαστε γιατί μετά την Ιταλία θέλουμε να αλλάξουμε από την κορυφή προς τα κάτω ολόκληρη την Ευρώπη και θα το κάνουμε με τη συνένεση του Ιταλικού λαού στις ευρωεκλογές. Η Λέγκα του Σαλβίνη θα γίνει το πρώτο κόμμα της Ιταλίας και το πρώτο κόμμα ολόκληρης της Ευρώπης. Ε, δεν θα είμαστε σκλάβοι των τραπεζών και των πολιεθνικών, των σπρέντ και της λιτότητας. Τέλος στην Ευρώπη του Γιούνκερ, της Μέρκελ και του Μακρόν που θέλουν να ταπεινώνουν τους λαούς και το λαό της Ιταλίας. Στην Ιταλία το λόγο έχουν οι Ιταλοί πολίτες, όχι η Μέρκελ ή ο Μακρόν. Μετά τις ευρωεκλογές θα έχουμε την δύναμη να δημιουργήσουμε μια νέα Ευρώπη, την Ευρώπη των λαών της ελευθερίας, της υπεράσπισης των συνόρων, τη, του Made in Italy, της αναχέτησης των μεταναστών στα σύνορά μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζουμε ότι η κυβέρνησή μας θα διαρκέσει για πολύ, θα είναι για πολύ στην εξουσία, γιατί έχουμε μία αποστολή να υπερασπιστούμε τη γη μας από τους γραφειοκράτες των Βρυξελών και να υπερασπιστούμε την εθνική κυριαρχία. Μπράβο σας κύριε Πρωθυπουργέ. Γουλφ από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε Πρωθυπουργέ Κόντε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σήμερα. Κύριε Πρωθυπουργέ της Ιταλίας, η αποφασιστικότητα της κυβέρνησής σας να αντισταθεί στη, στα, στην προνομιακή πρόσβαση στην εξουσία της Μέρκελ και του Μακρόν και να αντισταθεί στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελίτ που είναι εδώ παρούσες και προτείνουν ότι η κυβέρνησή σας είναι ρατσιστική, φασιστική και ότι είναι ανδρίκελα του Πούτιν και ότι είναι αντιφεμινιστική και αντιευρωπαϊκή. Σας χειροκροτώ για την δράση σας. Εσείς εμπνέετε τους δημοκράτες παντού στην Ήπειρο και στον κόσμο. Η κυβέρνησή σας έχει καταδείξει ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτός ο θεσμός που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είναι ένας, ε, μία ήπειρος αρχαίων λαών, αρχαίων εθνών. Αρχαίων λαών, αλλά με σύγχρονες μεθόδους. Ορισμένες φορές φοράνε κίτρινα γυλαίκα. Ορισμένες φορές ψηφίζουν Brexit. Ορισμένες, όπως οι συνάδελφοί σας από τα πέντε αστέρια, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα και τα κάνουν πολιτική εξουσία για τους ε, απλούς ανθρώπους. Είναι σύγχρονες οι μέθοδοι για αρχαίες φωνές, αλλά οι φωνές αυτές πρέπει να εισακουστούν. Η συζήτηση σήμερα αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς και η κυβέρνησή σας και οι συναδελφοί σας είστε το μέλλον της Ευρώπης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στον Πρωθυπουργό της Ιταλικής Δημοκρατίας για να απαντήσει στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Μετά έχουμε το Catch the Eye. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα θέματα που θίξατε είναι ποικίλα κινούμαστε από θέματα ευρωπαϊκού αποτυπώματος σε θέματα που αφορούν την εθνική μας πολιτική, την πολιτική της Ιταλικής Δημοκρατίας. Θα αρχίσω από ένα θέμα που θίξατε, θα ομαδοποιήσω στις απαντήσεις μου και θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα που απασχόλησε σχεδόν όλους, ε, την μετανάστευση. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι αυτό που έκανε η κυβέρνησή μου συγκεκριμένα ήταν να δει την πραγματικότητα κατάματα. Ο καθένας μπορεί να αντλήσει τα συμπεράσματά του, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα γεγονότα αυτά. Από την πρώτη στιγμή αυτής της ε, πολιορκίας γνωρίζουμε βέβαια ότι η μετανάστευση οδηγεί σε διχογνωμίες και τη στιγμή που είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες ελιμενισμούς δεν είχαμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές γιατί λόγω της γεωγραφικής μας ε, θέσης, μερικοί το ξεχνάτε, αλλά είμαστε στην καρδιά της Μεσογείου και από την ε, κεντρική Αφρική έχουμε άπειρες ροές. Γνωρίζοντας το τι συνέβη και γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτή μία αλόγιστη υποδοχή γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να υπάρχει και ένταξη. Δεν γίνεται ένταξη έτσι. Ένα συνάδελφός μου, ένας πρωθυπουργός ευρωπαϊκής χώρας, είχε αντιμετωπίσει την μετανάστευση από απόσταση. Μετά μου είπε Τζουζέπε, κατανοώ ότι έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα όταν έβλεπα στους δρόμους ε, δεκάδες δεκάδες μετανάστες. Πώς το αντιμετωπίσαμε με μία διαρθρωμένη απάντηση. Καταλάβαμε ότι πρόκειται για μία κατεπίγουσα κατάσταση που δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε εύκολα. Ορίσαμε λοιπόν 10 στόχους σε σχέση με την πολιτική, ε, με τις χώρες διαμετακόμισης, από που αρχίζει αυτή η πορεία των μεταναστών, οι χώρες ε, διαμετακόμισης και εδώ μιλώ και για παράκτιες ε, χώρες. Μιλήσαμε λοιπόν για κατανομή αντιμετώπιση και επαναπατρισμούς. Κατά το πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Ιουνίου, όπου συμμετείχα, μιλήσαμε για αυτά τα συμπεράσματα, φτάσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα και μιλήσαμε για κοινές στοχοθετήσεις και όποιος στην στην ουσία φτάνει στην Ιταλία, φτάνει στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα το οποίο δεχτήκαμε. Έμπρακτα όμως, ακόμα και σήμερα, δεν έχουν βρεθεί λύσεις. Είχαμε πολλά ευρωπαϊκά συμβούλια έκτοτε, αλλά καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να θέσουμε σε εφαρμογή αυτές τις αρχές. Και δεν φταίει η Ιταλία γι' αυτό. Δεν φταίει η Ιταλία. Η Ιταλία φυσικά έσωσε την Ευρώπη στο παρελθόν και την τιμή της Ευρώπης. Αλλά δεν λύνουμε έτσι το ζήτημα υπερασπιζόμενη την τιμή της Ευρώπης. Γιατί όποιο κράτος βρεθεί στη δινή θέση της Ιταλίας φτάνει σε ένα σημείο κορεσμού. Οι μηχανισμοί ένταξης δεν λειτουργούν πλέον. Οι επαναπατρισμοί είναι δύσκολοι γιατί δεν είναι αποδοτικοί. Δυστυχώς με ορισμένες χώρες δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τους μετανάστες. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο διμερός πολλές φορές. Άρα, αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει ούτε επαναπατρισμός. Γι' αυτό φτάσαμε σε μια πιο αυστηρή στάση. Το λέμε. Το λέμε ανοιχτά. Με σαφήνεια και διαφάνεια. Γιατί θεωρήσαμε, αφού καταρτήσαμε αυτή τη διαρθρωμένη στρατηγική, ότι δεν μπορεί να γίνει πάγια τακτική. Δεν είναι ο μόνος δρόμος, αλλά ένας δρόμος για να σταματήσουμε την διακίνηση ανθρώπων. Υπάρχει μεγάλη υποκρισία στην Ευρώπη. Οι μετανάστες γίνονται πρόβλημα όταν τους βλέπουμε με τους προβολείς στη Μεσόγειο, όταν μίκιο το κάνει θέμα στα ΜΜΕ. Αλλά μην ξεχνάμε τους μετανάστες εκεί όπου άφησαν το χωριό τους και όπου τους αναλαμβάνουν οι διακινητές. Ξέρετε πόσο στοιχίζει αυτή η, πο, πορεία της ελπίδας μετά από βασανισμούς, μετά από μεγάλα βασανιστήρια, 3.500 δολάρια το ελάχιστο. Μιλάμε για φτωχούς ανθρώπους που έχουν μεγάλη δυσκολία να βρουν αυτά τα χρήματα και στη συνέχεια τους αποσπώνται και αντιμετωπίσουν μύρια όσα δεινά. Η Ιταλία μέσα στα πλαίσια του Search and Rescue σε αυτή τη διαδικασία διάσωσης προσπάθησε πάντα να τηρήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ισχύει και στην περίπτωση Ντιτσότη, γιατί είδαμε τους πιο ευάλωτους, τους ε, πήραμε και τους μεταφέραμε στη γη. Όπως και στην τελευταία περίπτωση είχαμε ένα πλοίο όπου ζητήθηκε η υγειονομική περίθαλψη, είδη διατροφής και μετά από ημέρες στο λιμάνι προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κακή μεταχείριση, αλλά φτάσαμε σε κοινά συμπεράσματα σε επίπεδο 28 και δεν μπορείτε ε, να λέτε ότι υπάρχει μηχανισμός επανακατανομής. Δεν λειτουργεί έμπρακτα αυτός ο μηχανισμός. Δεν είναι υποχρεωτικός για όλους. Ας φτάσουμε και σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Υπάρχει ασφαλές λιμάνι μόνο όταν αποβιβάζεται κανείς στην Ιταλία, μα δεν είναι το πιο κοντινό λιμάνι, το πιο σίγουρο. Ο μηχανισμός επανακατανομής δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο σε τρεις, τέσσερις, πέντε χώρες. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι σε αυτό το μηχανισμό αλληλεγγύης. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα. Μην το κρύβουμε. Υπάρχουν χώρες που λένε ότι είναι ε, διαθέσιμες να συμμετάσχουν στο μηχανισμό επανακατανομής, αλλά το κάνουν μόνο για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασίες. Κανένας δεν θέλει τους οικονομικούς μετανάστες. Παραμένουν στα λιμάνια αποβίβασης. Τώρα, για την οικονομία και για τις επενδύσεις και τις υποδομές, είπατε ότι η Ιταλία δεν θέλει να κάνει τις σωστές μεταρρυθμίσεις. Καλύτερα να πληροφορηθείτε γι' αυτό, γιατί στη διαδικασία διαμεσολάβησης με τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον αντιπρόεδρο, τους αντιπροέδρους ε, Ντομπρόφσκης και Μοσκοβισή από την πρώτη φορά που τους συνάντησα. Δεν τους είπα να μην μπούμε στη διαδικασία επί παραβάση. Τους έδωσα ένα κόρπους όπου αναφέρονται όλες οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει. Και είπαμε ότι η Ιταλία και είπαμε ότι δεν ισχύει ότι η Ιταλία δεν θέλει να κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε εγκρίνει και υλοποιούμε ένα ογκοδέστατο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων ε, περισσότερο από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Παρακαλώ, κατά την ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει θα κάνετε τις ερωτήσεις σας. Εγκρίναμε νόμο κατά της διαφθοράς που προβλέπει πρότυπα ε, κατά της διαφθοράς από τα πιο απαιτητικά, όχι μόνο στην Ευρώπη. Κύριε Ντάντε, αν θέλετε να μιλήσετε μετά, μετά. Μην διακόπτετε τώρα, παρακαλώ, φωνάζοντας. Παρακαλώ. Δεν μπορεί να γίνεται διάλογος μονομερής με το χρόνο που χάνουμε με τι διακοπέ δεν θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτέ. Προσπαθώ να απαντήσω. Θα, απαντήσετε μετά, θα απαντηθούν μετά οι ερωτήσει. Με τα απαιτητικότερα λοιπόν πρότυπα κατά τη διαφθορά, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά διεθνώ, έχουμε προβλέψει μια μεταρρύθμιση ρίζοσπαστική για την περίπτωση τη πτώχευση. Στην ε, Ιταλία δεν ε, γίνεται πια λόγο για πτώχευση ε, γίνεται λόγος για κώδικα των ε, εταιριών που χρειάζονται διάσωση. Μιλάμε για ένα ογκοδέστατο σώμα άρθρων. Θα πρέπει εδώ να δούμε τα σχετικά διατάγματα που χρειάζονται, τα νομοθετικά διατάγματα, για να απλοποιήσουμε όλες τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά. Πρέπει να γίνουν πιο ε, ταχείες οι όλες διαδικασίες. Αυτό έχουμε αρχίσει να το επιδιώκουμε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε καταξοδότηση πράξη και θα κοιτάξουμε να γίνει ροζοσπαστική ε, μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για τους δημόσιους διαγωνισμούς, τις προμήθειες. Έχουμε και άλλον νόμο για τον αστικό κώδικα, για την ε, εκδίκαση των υποθέσεων στα ποινικά δικαστήρια. Αυτά κάνουμε. Όταν λέτε ότι είμαστε κατά των επενδύσεων, μα τι να πω, παρακολουθείτε άλλες συζητήσει. ακούτε να μιλάνε άλλοι. Ε, με συγχωρείτε, αλλά το πρόγραμμα για τις επενδύσεις στις υποδομές στην Ιταλία. Το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει τις τεράστα, τα τεράστια κονδύλια που προβλέπονται για τις επενδύσεις, τα 13 δις πέραν των κρατικών επιχειρήσεων, οι οποίες όπως λέτε ε, έχουν έρθει παρόλα αυτά να συζητήσουν μαζί μας στο Μέγαρο Εδώ λοιπόν κοιτάζουμε ένα πρόγραμμα ασφάλειας για όλη τη χώρα ένα εθνικό πρόγραμμα για, τις, για τους κινδύνους υδρολογικού χαρακτήρα. Κοιτάζουμε να προστατεύσουμε τις, υδάτινες, τις υποδομές μας για την υδροδότηση. Και εδώ χρειαζόμαστε και ευελιξία. Το, το συναντηθήκαμε με την Επιτροπή και το αποσπάσαμε. 3 δις. 3 δις 200 εκατομμύρια επιπλέον πέραν του επενδυτικού προγράμματος που ήδη έχει οριστεί χρειαζόμαστε. Πρέπει να ακούσουμε και τις διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να υπάρχει διαφορά απόψεων Στη δημοκρατία αυτό είναι το ωραίο, ότι υπάρχουν συζητήσει για τα κοινά δημοσίω, οπότε ακούγονται διαφορετικέ απόψει. Όμω το να αγνοεί κανεί όλα αυτά σημαίνει ότι ουσιαστικά ε, κοροϊδεύει του ε, Ευρωπαίου πολίτε, όχι μόνο του Ιταλού. Σε ό,τι αφορά την ΤΑΒ, Σε αφορά λοιπόν τα γρήγορα τρένα, είναι ένα πρόγραμμα που ήδη εγκρίθηκε. Ε, η κυβέρνηση ήδη θεωρεί ότι είναι ορθό απέναντι στις ανάγκες των πολιτών, ακριβώς επειδή επιπλέον υπάρχουν και αξιολογήσεις ε, που δικαιολογούν αυτό το έργο. Εδώ και 25 χρόνια υπάρχουν. Τώρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να υλοποιηθεί. Ε, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η προκαταρκτική φάση, αλλά πριν αρχίσουμε να εκτελούμε και να χρησιμοποιούμε, να ξοδεύουμε τόσα πολλά κονδύλια, πριν πραγματοποιηθούν τέτοιε υποδομέ που έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον, γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια ανάλυση ωφελία. Είπαμε ότι θα την κάνουμε με διαφάνεια. Όταν θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα, και ότι θα αναλάβουμε τις σχετικές ευθύνες για τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν. Σε ό,τι αφορά τα άλλα προγράμματα, όλα βρίσκονται στη φάση υλοποίησης. Ε, ο αυτοκινητόδρομος στο Μπρένερο, η ΤΑΠ και οι επιταχύνσεις στις επενδύσεις και στα των εργοταξίων θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, με ταχύτητα σε όλα τα σχετικά έργα. Και με συγχωρείτε, Πρόεδρε, που θα καταχραστώ το χρόνο σας, αλλά δύο κουβέντες και για την εξωτερική πολιτική. Μας λέτε πολιτική απομόνωση. Η Ιταλία λέει είναι σε πολιτική απομόνωση. Για την Βενεζουέλα εμπόδισε τη διαδικασία και παρέμεινε απομονωμένη. Προσοχή εδώ, προσοχή. Πάνω απ' όλα, η Ιταλία σε καμία περίπτωση δεν είναι απομονωμένη συνεισέφερε τα μάλα, και αυτό είναι γεγονός, στην έκδοση των ανακοινοθέντων από την ύπατη εκπρόσωπο. Στις 26 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις, ε, ε, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι και τη δική μου η τοποθέτηση ήταν η καθοριστική σημασία για να προκύψει αυτό το ανακοινοθέν. Πολλοί θέλουν να γράψουν την ιστορία πριν γίνει. Καλό θα ήταν εδώ να φανούμε συνετοί. Ε, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση στην κρίση της Βενεζουέλας. Η Ιταλία ξέρει πολύ καλά τι κάνει και δεν είναι η μόνη. Είναι πολλές άλλες οι χώρες που έχουν ξεκάθαρες απόψεις. Ξέρουμε τι γίνεται και το θυμίζω για μας οι προεδρικές εκλογές του 2018 στη Βενεζουέλα δεν ήταν δημοκρατικές εκλογές, δεν τις αναγνωρίσαμε. Ναι, και επίσης ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζονται νέες προεδρικές εκλογές στη χώρα. Χρειάζεται να γίνουν με συνθήκες νομιμότητας, με διαφάνεια, να είναι αξιόπιστες βάσει των διεθνών προτύπων. Τις θέλουμε όσο δυνατόν νωρίτερα. Ε, γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε πλήρη επίγνωση, ότι υπάρχει ένας μεγάλος ρυθμός πολιτών που υποφέρουν και ήδη έχουμε προβλέψει από τα κονδύλια για καταπήγουσε ανθρωπιστικές ανάγκες σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα να στείλουμε ποσά. Γνωρίζουμε ότι κανένα καθεστώς δεν μπορεί να δικαιολογεί την ύπαρξή του με τις βίες ενέργειες, με την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων με βία. Όμως θεωρούμε ότι δεν μπορούμε και να παρέμβουμε δεν μπορούμε να ε, ε, στέψουμε και να αναγνωρίσουμε κάποιον ο οποίος δεν προέκυψε ως αρχηγός ε, κράτους ή κυβέρνησης από ελεύθερες ανεξάρτητες εκλογές. Θέλουμε να δημιουργηθεί ομάδα επαφή, μια μορφή διαμεσολάβηση όπου να συμμετάσχουν όλοι. Υπάρχει ιστορική ευθύνη εδώ. Ιστορική ευθύνη να πούμε ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποιον, σε το αξίωμα ε, ει βάρο κάποιου άλλου. Φανταστείτε στι μεγαλύτερε διεθνεί κρίσει από ιστορική ε, σκοπιά ε, τι εξέλιξη θα είχαν αν δεν είχαν όλοι βιαστεί να αναγνωρίσουν κάποιον πρωταγωνιστή και σε είπα το αξίωμα ενώ υπήρχε ο αντίπαλός του ακόμα ε, στο προσκήνιο. Εδώ λοιπόν ριζοσπαστικοποιείται η αντιπαράθεση. Το να αναγνωρίσει κάποιο τον ένα σημαίνει ότι υποχρεώνει του διεθνεί πρωταγωνιστέ στα διεθνή πράγματα να πάρουν το μέρο του άλλου. Θα γίνει χειρότερη κρίση σε σχέση με αυτέ που σέρνονται ακόμα στι σελίδε τη ιστορία μα. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη συζήτηση με τη διαδικασία Catch the Eye. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το πολύ στις 19 και 45. 50 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Όσο περισσότερο μιλάτε εσείς, τόσο λιγότερο θα μιλάνε οι άλλοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, Υπουργέ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλήσατε για δημοκρατία. Εδώ πέρα βρίσκεστε ίσως στο πιο δημοκρατικό θεσμικό όργανο, γιατί είμαστε αμέσως έρετοι από τους ε, πολίτες. Σε αντίθεση με εσάς ε, που διοριστήκατε. Εγώ είμαι περήφανη που είμαι Ιταλίδα, είμαι στο πλευρό της Ιταλίας, αλλά της Ιταλίας στην Ευρώπη. Και κοιτάξτε, ε, μας είπατε ότι υπάρχει ακριβώς ε, το θα είναι περίπατος ε, το θέμα αυτό του Made in Italy, μεταρρύθμιση του Δουβλίνου κτλ. Ότι μας λέτε εργαστήκατε και έχετε κάνει συμμαχίες, συμμαχίες που δεν υπάρχουν στην Ιταλία, συμμαχίε που δεν υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μιλάτε για την Ευρώπη, μιλάτε για ενότητα και μετά μας λέτε ότι δεν θα κάνετε το τρένο, το TAV. Δεν ξέρω αν ε, κάνω λάθος. Μετά μιλάτε για μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και ακούμε συνεχώς ότι τα πράγματα αυτά θα γίνουν προαιρετικά. Μα ε, τι αλληλεγγύη ε, μιλάμε μετά και τι αλληλεγγύη ζητάτε όταν θέλετε να είναι προαιρετικά. Είναι λοιπόν δικό σας το λάθος και καταλήγω. Το βίντεο σας με την καγκελάριο Μέρκελ είναι ντροπή γιατί εγώ αγαπάω την Ιταλία και δεν θέλω να κακολογεί ε, ο Πρωθυπουργό στην Ιταλική κυβέρνηση σε μια ομολογό του. Σας ευχαριστώ, Γκυγιόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε τη Κυβέρνηση, όταν δεν είμαι στο Στρασβούργο και τι Βρυξέλλε, ζω στη Λιόν. Είναι μια πόλη που έχει αρχαίου δεσμού με την Ιταλία. Είναι πολύ κοντά στο Πιεμόντε και βεβαίω το 16ο αιώνα ήταν πολλοί Λιονέζοι που μετανάστευσαν στην Ιταλία και αντιστρόφω πολλοί Ιταλοί μετανάστευσαν σε εμά. Και στο Τωρίνο, ε, τον αυτοκινητόδρομο που θέλουμε να φτιάξουμε Τωρίνο Λιόν, πώ γίνεται ακόμα να είναι στα χαρτιά. Δεν είναι απλώ για να συνδέσουμε δύο πόλει, είναι γιατί και το καλύτερο λέει από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει ένα δρόμο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το θέμα τη λεκάνη τη Μεσογείου και την διασύνδεση ε, μεγάλων πόλεων μεταξύ του. Μιλάμε λοιπόν για δεσμού. Ε, υπολογίζουν όλοι τα λεφτά, έχουν κάνει οι λογιστέ του απαραίτητου υπολογισμού και έχουν δει τι θα κοστίσει αυτό στο Ιταλικό κράτο. Σίγουρα σε πρώτη φάση τα έσοδα θα είναι λιγότερα από τα έξοδα και θα υπάρχουν οι φόροι του καυσίμων, λιγότερε οδικέ μεταφορέ, λιγότερα φορτηγά, λιγότερη ρήπανση. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξή. Δεν πιστεύετε ότι ο αδερφικό και παλιό δεσμό που ενώνει τι δύο χώρε μα δεν πρέπει να πάρει και πολιτική έκφραση, ε, ώστε να μην εμποδιστεί από ιδεολογικέ περιβαλλοντικές μέρημνε. Ευχαριστούμε κύριο Κύριε Πρωθυπουργέ, σα ευχαριστώ για τι δηλώσει σα. Μίλησατε πολύ για αλληλεγγύη που ζητάει τώρα η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η συνεισφορά σα αυτή στο μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ζητάτε ε, αλληλεγγύη. Αλλά όταν μιλάμε για αλληλεγγύη πρέπει να μιλήσουμε και το γιατί καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση όπου αναγκάζει την Ιταλία να ζητήσει αλληλεγγύη. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από 20 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια έχουμε ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ. Και εδώ και 15 χρόνια η Ιταλία δεν έχει καμία ανάπτυξη. Έχετε σκεφτεί μήπως υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δύο. Μήπως η Ιταλία θα έπρεπε να σκεφτεί αν κάνει αυτό το νόμισμα για τη χώρα θα μπορούσε, δεν ξέρω, η Ιταλία διαφορετικά να δημιουργήσει ένα έλλειμμα target 400 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μήπως οφείλεται εκεί στο ότι η Ιταλία συνεχώς παραβιάζει τους κανόνες ε, για το έλλειμμα. Κύριε Κόντε, όταν ζητάτε αλληλεγγύη πρέπει να τηρεί και τους κανόνες η Ιταλία. Στο σύστημα του ασύλου δεν το κάνετε. Πρώτα απ' όλα δεν τους καταγράφετε όλους και τώρα κλείνετε όλα τα λιμάνια και έχετε πάει στο άλλο άκρο. Λοιπόν, αν θέλει να είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Ιταλία, πρέπει να τηρεί του ευρωπαϊκού κανόνε. Αλλιώ δεν μπορεί να υπάρξει αλληλεγγύη. Σα ευχαριστώ. Τάραντ. Ονορεύει Μιράντα. Μιράντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ Κόντε, γιατί εμπόδισε η κυβέρνησή σας ένα σκάφος διάσωσης να ελιμενιστεί το 2018. Εγώ με τέσσερις ευρωβουλευτές του Κοινοβουλίου ε, επισκέφθηκα την Ιταλία και δεν πήραμε επίσημη απάντηση. Ο Υπουργό Μεταφορών σα είπε ότι πρόκειται για θέματα δημοσία τάξη και τέτοιου λόγου που εμπόδισαν τον ελληνισμό. Ε, οι εκπρόσωποι τη Ιταλική κυβέρνηση ε, δεν μπορούσαν να μα εξηγήσουν γιατί έκτοτε μπλοκάρονται τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Γιατί μιλάτε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όταν δεν σέβεστε του κανόνε. Κανόνε αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, σοκάρει το γεγονό ότι από στόματο τη ε, επίσημη κυβέρνηση, που θα μπορούσε να είναι πιο δημοκρατική, υπάρχουν διασυνδέσει με την ακροδεξιά, με φίλου του φασισμού, με φίλου όσων είναι αντίθετα με όσα προσβεύει η Ευρώπη. Ε, ο κύριο Μποργκέτσου. Στο νέο αρχηγό της κυβέρνησης, Πρέπει να πω ότι προσφέρεται και πάλι αξιοπρέπεια σε μια χώρα που δεν ήταν συνηθισμένη σε αυτό. Ε, ένα λαό που, δεν είχε, συνηθί, που είχε συνηθίσει μάλλον να βλέπει ε, κολλημένου στον τοίχο του εκπροσώπου του όταν έρχονταν στην Ευρώπη. Καταφέρατε να πετύχετε πολλά ενώ υπήρχε η τάση ρήξη σε μια χώρα, σε μια χώρα καταφέρατε να, ε, να δείξετε ανάγλυφα την αλήθεια, την αλήθεια των γεγονότων, ότι η χώρα μας είναι μια μεγάλη χώρα όπου όλοι δουλεύουν σκληρά και ότι είναι σημαντικό να υπάρχει χρηματοδότηση, να στηριχθεί η οικονομία. Ζηλεύουν οι άλλες χώρες, ζηλοφθονία υπάρχει και πολλές φορές έχουν εκβιάσει ε, με, τις πολιτικές, με τα πολιτικά τους προσχήματα, προσπαθούν να περάσουν πολιτικούς στόχους και ευρωπαϊκούς, η οποία όμως είναι ουσιαστικά απόρρια χειραγώγησης. Σας ευχαριστώ λοιπόν που δείξατε τέτοια ε, σταθερότητα και στη συνεργασία με την άλλη συνιστόσα της κυβέρνησής σας που θέλει ε, να δείξει ότι η Ευρώπη είναι αρκετά απρόσεκτη, ότι το γεγονός ότι δεν καταφέρνει να εμποδίσει το εμπόριο ανθρώπων στην Μεσόγειο είναι ψεύδος και εξυπηρετεί άλλους σκοτεινούς σκοπούς. Η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, το εμπόριο αυτό εμποδίστηκε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την προσπάθεια που αναφέρατε να γίνει άνοιγμα προς τις αφρικανικές χώρες με τις οποίες πρέπει να υπάρξει διάλογος, να υπάρξουν συνθήκες αξιοπρέπειας και ισοτιμίας και εκεί και σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια ανοίγματο και συμμετοχή στο σύστημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας, στην υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο διότι μόνο σπήροντας έναν υγιή σπόρο, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πρόσφορο έδαφος, τότε θα προχωρήσουμε. Όχι αυτά που κάναν οι παλιοί κυβερνώντες που πήγαιναν και άπλαναν τα πλοκάμια του στην Αφρική και κλέβαν από την Αφρική. Αυτό πρέπει να κάνει ένας αξιοπρεπής τίμιος λαός. Ευχαριστούμε κύριε Μποργκέτσι, ο κύριο Βόιτ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε. Καταφέρατε να σταματήσετε αυτή την μαζική εισβολή μέσω της Μεσογείου. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Δεν είναι μυστικό ότι το λόμπι του ασύλου πλέον βγάζει λιγότερα λεφτά από ό,τι στο παρελθόν και το καταφέρατε εσείς. Και γι' αυτό κάνουν σαν να σας δικάζουν σήμερα. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι δικαστήριο. Τρίζουν οι παλιές ελίτ γιατί ξέρουν ότι σε τρεις μήνες δεν θα είναι πια η πλειοψηφία εδώ μέσα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, στη Γερμανία είδαμε ότι μπορούν και να σκοτώσουν οι μετανάστες κατά χιλιάδες. Σταματήστε τους φόνους και δώστε στα εκατομμύρια Ευρωπαίους που κοιτάνε σήμερα προς την Ιταλία και την Πολωνία την ελπίδα για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Χιμένες Πεσερίλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμερίζομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, αναχαιτήσουμε και να καταπολεμήσουμε το εμπόριο ανθρώπων στην Αφρική. Όμω δεν συμμερίζομαι την ουδετερότητα, τη στάση ουδετερότητα τη Ιταλία για το θέμα τη Βενεζουέλα. Διότι μπλοκάρατε την αναγνώριση του Γκουαϊντό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ την έχω την Ιταλία στην καρδιά μου. Έχω ε, παιδιά που είναι Ιταλοί στην εθνικότητα, στην Ιθαγένεια. Έχω ζήσει εκεί πάνω από 20 χρόνια και δεν καταλαβαίνω πως ένας Ιταλός δεν βλέπει την κατεπίγουσα ανάγκη ε, της... Ε, απομάκρυνση του κυρίου Μαντούρο που καταστέλει τα δικαιώματα των ε, κατοίκων τη Βενεζουέλα. Μιλήστε με τον κύριο Λόπε, μιλήστε με όλου του βασανισμένου, αυτού που έχουν βρεθεί στον τάφο, όλου αυτού του μετανάστε που βρίσκονται εκεί ε, και ζουν σε ένα φέρετρο στην ε, Κολομβία. Όπω είπε κάποιο, το μόνο απαραίτητο για να σταματήσει το κακό είναι να παραμένουμε αδρανείς. Είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος. Αναφέρομαι, ε, σας απευθύνομαι ως πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Στην ε, περιφέρεια μου παίρνουμε πολλά ε, εκατομμύρια ευρώ για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ιταλία για την παράκτεια και ορεινή όμως δράση μας. Δεν γίνεται τίποτα από την πλευρά της Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή θα σας θυμίσω την ανάκληση του πρέσβη σας, ε, του πρέσβη μας μάλλον από τη χώρα σας και ότι πρέπει να υποστηριχθούν ξανά οι σχέσεις μας. Πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες διπλωματικές προσπάθειες που να δείχνουν ότι τα λόγια σας είναι πραγματικά υπέρ της Ευρώπης. Ε, στην ε, Γαλλία δείχνουν, φαίνεται ότι η πολιτική που χαράσουμε δεν μπορεί να συνδυαστεί με τη δική σας που απλώς μιλάει υπέρ της εθνικής κυριαρχίας της Ιταλίας και δεν έχει στόχο να είναι αποτελεσματική. Εάν θέλετε να υποστηριχθούν οι Ιταλοί φορολογούμε μόνο, θα αυτό θα είναι ει βάρο των Γάλλων πολιτών όμω και των Γάλλων ψηφοφόρων. Μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει προεκλογική εκστρατεία και ηθικέ ευθύνε. Με ένα φίλο σαν και εσά, τι να, κάνει, τι να κάνει κανεί του εχθρού. Η συμπεριφορά σα είναι άκομψη, αγενή, αφθάδη, ε, παράνομη και ε, συμμορήτικη. Θα πρέπει λοιπόν να ε, σα πω ότι δεν σα απευθύνω καμία αναγνώριση γιατί δεν σα αξίζει. Κυρία Τόγια. Ε, Πρωθυπουργέ, από τα λόγια των συναδέλφων εδώ ακούγεται πόση σεβασμός και εκτίμηση υπάρχει για την Ιταλία και πόση απογοήτευση και ανησυχία των φίλων μας για την Ιταλία. Πρέπει να τη δούμε πιο αντικειμενικά. Έχει αποδυναμωθεί, έχει απομονωθεί. Ε, υπάρχει διένεξη με τους συνεργάτες με τους οποίους θα πρέπει να χτίζουμε ένα κοινό μέλλον. Πώς μπορεί να είμαστε κατά της Ένωσης και της αλληλεγγύης. Εσείς τα είπατε, μόνο σας. Θα πρέπει λοιπόν με ευφυΐα και ε, να, να ε, ε, αρπάξουμε αυτή τη ευκαιρία. Και το λέω με απογοήτευση και όχι με χαρά, γιατί θέλω η Ιταλία, η χώρα μου, να είναι πρωταγωνίστρια στι μελλοντικέ εξελίξει. Και κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να ξεφύγουμε από τα πατηλά όνειρα και τι μεγάλες, ε, ε, ε, τα μεγάλα οράματα και τις χήμερες για το τι θα γίνει στη Μεσόγειο. Εδώ πρέπει να αλλάξει η στάση μας. Πού είναι η συνοχή για την οποία μιλάτε. Θα σας πω δύο πράγματα. Δεν λέω ότι τα καταφέραμε εμείς, γιατί η Ιταλία δεν φεύγει τώρα από την Ευρώπη αλλά να σα θυμίσω τα εξή και πείτε μου αν αυτή η εξοπιστία είναι ευρωπαϊκή, κύριε Πρωθυπουργέ. Για το κονδύλι για την Αφρική, η πλειοψηφία σα ψήφισε κατά. Ε, για τα δισεκατομμύρια του προγράμματο Juncker, τα δικά σα κόμματα που τώρα ε, κυβερνούν ε, ψήφισαν κατά. Για την απέτηση τη ενισχυμένη συνεργασία, γιατί η Ιταλία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία των 9. Κατά. Για τι αρνητικέ συνέπειε του Brexit. Δεν ξέρετε ότι το μεγαλύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ιταλία είναι αυτό του Φάραντ μέσα από το δικό σα στο ε, διάβλο. Ε, κυρία Τόγια, κυρία Τόγια, παρακαλώ. Σα παρακαλώ λοιπόν να τρέψετε στην Ιταλία να ξαναγυρίσετε στη σωστή τροχιά. Ευχαριστούμε ο κύριο Ρανζέλη. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, προφανώς ε, με, το λόγο σας που ακούσαμε εδώ και με την τεράστιο σεβασμό που σας απευθύνουμε πρέπει να πω τα εξής. Ένα σημείο θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ θα πρέπει να θυμίσω τον Άλτο Μόρο και να θυμίσω ότι η τωρινή κυβέρνηση τη, ε, δεν θα πρέπει να θάψει τη μνήμη του Μόρο και την φιλευρωπαϊκή του στάση. Δεν αρκεί όμω να τον αναφέρουμε σε σχέση με τη Μεσόγειο, πρέπει να τον αναφέρουμε και σε σχέση με την Ευρώπη. Ε, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι ω Πορτου... Πορτογάλο ευνηδιάζομαι από τη στάση τη Ιταλική κυβέρνηση στα θέματα τη Βενεζουέλα. Όχι απλώ γιατί θέτει ένα αμφιβόλο το όλο θέμα τη ευρωπαϊκή εξωτερική δράση, αλλά γιατί υπάρχει πορτογαλική κοινότητα στο Καράκα, στη Βενεζουέλα και υπάρχει και μεγάλη κοινότητα Ιταλών. Η Ιταλική κυβέρνηση δεν σκέφτεται του Ιταλού που ζουν και υποφέρουν λόγω του καθεστώτο του Μαδουρό, γιατί έχουν να υποστούν τα βασανιστήρια που του επιβάλλουν αυτή είναι η ερώτησή μου προ την Ιταλική κυβέρνηση. Ήδη θα έπρεπε να είχατε τοποθετηθεί. Δεν αρκεί να απαντήσετε τώρα. Έπρεπε να έχετε απαντήσει στην πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη. Μικρόφωνο. Έχω μια ερώτηση κύριε Πρωθυπουργέ. Πώς ε, βλέπετε ότι θα γίνει η κοινότητα, μια κοινότητα αλληλεγγύης ε, στα θέματα της ε, μετανάστευσης, πώς είναι δυνατόν να μας πηγαίνετε προς μια κατεύθυνση που, που επευλήθηκε στη Γερμανία με τους νόμους Χάρτς 4. Πώς είναι δυνατόν να σας επιβάλλουν τα πέντε αστέρια την ατζέντα τους στα κρίσιμα ζητήματα. Και είναι σοβαρά αυτά τα ερωτήματα, γιατί ακριβώς τη στιγμή που η Λέγκα αγκαλιάζει τις δυνάμεις της άκρας δεξιάς που θέλουν να πέσει η κυβέρνηση, μιλάτε ακριβώς για αλλαγή καθόλου στην ε, Βενεζουέλα. Λοιπόν, σε τι βασίζεστε ως πρόβλεψη και ως ε, μελέτη ότι φέτος και τα επόμενα χρόνια θα είναι θαυμάσια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα μια απάντηση. Ο κύριος Σαλίνη. Πρόεδρε, καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα φανώ πραγματιστή. Ε, θα ήθελα να έχω χρόνο για να περιγράψω τι ε, κόπο έχει προκαλείται, ε, μάλλον με τι κόπο ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καταφέρουν να αποσπάσουν εκατομμύρια κονδύλια για τα έργα και τα προγράμματα που εκτελούνται στι διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε, μεταξύ των οποίων η δική μου. Θα χρειαζόμουν πολύ χρόνο για να αφηγηθώ πώ προσπαθήσαμε μέσα στο πέρασμα του χρόνου να δημιουργήσουμε σοβαρά προγράμματα που να συνδυάζουν τι απαιτήσει διασύνδεση τη χώρα μα τι απαιτήσει των επιχειρηματιών μα. Θα ήθελα να τα θυμίσω όλα αυτά και να αφηγηθώ κιόλα ε, σε τι ψυχική κατάσταση βρίσκονται όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ο ίδιο Υπουργό των Υποδομών και ότι ασχολείται περισσότερο με τις ε, χημικές ε, με τα χημικά απόβλητα παρά με αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν ο, η κυβέρνησή σα να μας αποδείξει τι τεράστιε δυνατότητέ τη, τι οποίες διαφημίζετε. Εγώ θα σας προκαλέσω στο εξή. Ε, πολλοί ε, έχουν, προκαλέσει το, έχουν απευθύνει προκλήσεις ε, σε κυβερνήσεις για πολιτικού σκοπού με αντικείμενο του μισθού. Εάν θέλετε λοιπόν να κάνετε μια αλλαγή στη χώρα, προβλέψτε ένα αντασφαλιστικό δάνειο ε, με σταθερό επιτόκιο και επιστρέψτε από τη δική σας την τσέπη για να δούμε πώς θα γεμίσουν τα ταμεία της χώρας μας. Ευχαριστούμε ο κύριος Βιώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρωθυπουργέ Κόντε, θα σας πω κάποια, κάποιους αριθμούς που είναι βαρετά ίσως 2 στα 6, 3 στα 4 για τον Σαλβίνη ε, ψηφοφορία λοιπόν. Ε, αποτελέσματα ψηφοφοριών ήταν αυτό και αυτές είναι οι απουσίες των Υπουργών της Ιταλίας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για νέους, μιλάμε για μηχανία, για μεταφορές, για μετανάστευση. Δεν είστε εκεί. Δεν είστε στι συνεδριάσει του Υπουργικού Συμβουλίου. Ζητήστε συγγνώμη από του Ιταλού. Ζητήστε συγγνώμη από από του πολίτε τη Ιταλία και τη Ευρώπη. Δεν είναι αυτό η Ιταλία. Η Ιταλία χρειάζεται κυβέρνηση που να είναι παρούσα στην Ευρώπη. Να τη χρειαζόμαστε. Αυτέ τι δικαιολογίε που μα λέτε σήμερα, Πρόεδρε Κόντε, θέλουμε να ακούσουμε. Θέλουμε να είστε παρόντε πάνω απ' όλα και να κλείσουμε ένα παράθεμα. Ε, το είπατε κι εσεί, Πρόεδρε από το τραγούδι που κέρδισε το φεστιβάλ του Σαρέμο, του Μαμούτ. Ε, ότι είναι δύσκολο κανείς να αλλάξει τον κόσμο αν δεν έχει καμία περηφάνεια. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η Ιταλία ε, δεν έχει πια τίποτα για το οποίο να είναι περήφανη. Κοιτάξτε πώς είναι αδιαίθουσα. Παρακαλώ να χρησιμοποιείτε γλώσσα δέουσα και πρέπουσα για την Σύνοδο της Ολομέλειας. Ιδάλλως θα προβλέψω κυρώσεις για του βουλευτέ που χρησιμοποιούν ε, διατυπώσει που δεν είναι κόσμιε και δεν αρμόζουν στο χώρο του Κοινοβουλίου. Δεν θα το ξαναπώ. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρωθυπουργέ της Ιταλίας, κύριε Κόντε, Μεσχέ Κόντε, Σενιόρε Κόντε, αν μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά. Can I start from the beginning? Κύριε Κόντε, είμαι σύμφωνος με αυτά που λέτε για την πορεία της Ευρώπης. Αλλά η Ευρώπη πρέπει να δείξει αλληλεγγύη. Και η αλληλεγγύη πρέπει να εκφραστεί και στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, στον τομέα της ασφάλειας. Και γνωρίζετε ότι η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα, συνεχίζει να απειλεί την Κύπρο παραβιάζει συνεχώς τον εναέριο χώρο της ελλάδος παραβιάζει τα χωρικά ύδατα της ελλάδος παραβιάζει την αοζ της κύπρου και θέλω μια δήλωση δική σας στήριξης της ελλάδος έναντι των απειλών της τουρκίας μια δήλωση δική σας που να στηρίζει την κύπρο να μπορεί να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους τη στιγμή μάλιστα που η ιταλική εταιρεία η eni θέλει και αυτή να αξιοποιήσει και να συνεργαστεί με την κύπρο για αξιοποίηση των φυσικών πόρων και απειλείται και η ιταλία και η Έννη και η κύπρος από την τουρκία. θέλουμε μια δήλωση δική σας εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στήριξης της ελλάδας και της κύπρου και καταδίκης των απειλών του ερντογάν και της τουρκίας κύριε πρωθυπουργέ. το περιμένει ο ελληνικός λαός το περιμένουν επίσης οι φίλοι μας στην κύπρο. θέλουμε δήλωση συμπαράστασης. Καλώ Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να μπορείτε να με ακούτε. Ε, ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ, που ήρθατε. Ήταν έκπληξη. Θετική να σας ακούω. Και όπως λέμε στην Ίστρια, ε, θα πρέπει να μην ε, πουλάμε θήκια για μεταξωτές κορδέλες, θέλουμε και γεγονότα. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε μια καλή συνεργασία και για την ιδιατρική. Με ενδιαφέρει να μου πείτε πώς βλέπετε τις σχέσεις με τη Σλοβενία και την Κροατία και πώς βλέπετε να διαμορφώνετε το μέλλον για την συνεργασία με την Αδριατική. Είναι σημαντικό να μου πείτε πώς βλέπετε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Και επίσης με ενδιαφέρει αν η κυβέρνησή σας θέλει να περικόψει κονδύλια για τις Ιταλικές μειονότητες, ε, για τη διγλωσία κύριε Υπουργέ. Ε, πρωθυπουργέ μάλλον, ε, για την οποία εργάστηκα εγώ με συναδέλφου μου, ε, για την διγλωσία στην Σλοβενία και την Κροατία. Χρειαζόμαστε χρηματοδόσει και από την Ιταλία, λέει ο μιλητή, στην Σλοβενία και την Κροατία. Θα μπορούσε να υπάρξει και ειδική σύνοδος που να ασχοληθεί με τα θέματα που αφορούν τους μετανάστες και τους ε, κατοίκους των άλλων χωρών. Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επενέσατε ε, και μιλήσατε για την σημασία τη ελεύθερη κυκλοφορία. Θα συμφωνήσω. Είμαστε η μεγαλύτερη γλωσσική μονότητα που ζει στην Ιταλία κοντά στα σύνορα. Όμως η κυβέρνησή σα ε, έχει προβλέψει νόμο, το λεγόμενο Διάταγμα για την Ασφάλεια, που έχει να κάνει με πολλά άλλα, κυρίω με τη μετανάστευση και δεν θέλω να το σχολιάσω. Όμω βάσει αυτού του διατάγματο, εάν ένα ή κάποιο που θέλει να εργαστεί στο εξωτερικό πάει στο εξωτερικό, αγοράσει ένα αμάξι και θέλει να γυρίσει στην Ιταλία, το αμάξι αυτό θα το, το κατασχέσουν στα σύνορα και θα πληρώσει και 500 ε, ευρώ πρόστιμο. Μπορείτε να μου πείτε ένα τέτοιο μέτρο συνάδει με το μεγάλο ιδεώδες της ελεύθερης κυκλοφορίας που προσπιστήκατε. Ευχαριστούμε κύριο Σταραμπέλα. Είμαι πολύ ε, χαρούμενο που μπορώ να σα απευθυνθώ σήμερα, διότι ο κύριο Σαλβίνη, ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνησή σα, που ήταν πριν από λίγο καιρό εδώ στο Κοινοβούλιο, μα είπε τι απόψει του για του πολίτε, αλλά μακριά από τι κάμερε. Ελεύθερα, λοιπόν. Θα Ήθελα να μου πείτε λοιπόν για αυτό τον τρόπο δράση ε, στην κυβέρνησή σα. Λίγα γίνονται και πολλά ε, ακούγονται ιδίω σε επίπεδο φιλιαρία. Επίση, πολύ εύκολα δακτυλοδεκτούνται οι ένοχοι για όσα σημαίνουν την Ιταλία. Πρόσφυγε, Αφρικανοί, ε, ομοφυλόφιλοι, Γάλλοι, η ίδια η Ευρώπη. Ε, κάποια στιγμή οι ένοχοι ήταν οι Εβραίοι και οι κομμουνιστέ, ή οι Τσιγκάνοι, Αθήγανοι. Είναι τρόπο αυτό ε, να κάνει κανεί πολιτική. Δεν θυμίζει το φασισμό. Ε, αυτός κατέστρεψε την Ιταλία. Ε, ανάγκασε ε, εκατομμύρια Ιταλούς μετά τον πόλεμο να μεταναστεύσουν για να ζητήσουν το μέλλον τους. Σας παρακαλώ, μην το λησμονείτε. Ο κύριος Τσίκου. Ε, Σας ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η χώρα, η μας περνάει μια φάση ύφεσης και δεν άκουσα κύριε Πρωθυπουργέ δυστυχώς να μιλήσετε για τη βιομηχανική πολιτική, την εμπορική πολιτική δεν άκουσα να μιλήσετε για τις επιχειρήσεις μας οι εμπορικές συμφωνίες ε, που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σημαίνουν ε, ε εξαγωγές, εισαγωγές και ανάπτυξη θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί η φορολογία για να μπορέσουν να δώσουν δουλειέ οι επιχειρήσει μα και να, να σταματήσουμε τι επιδοτήσει που δεν χρησιμεύουν ε, σε τίποτα παρά να παριστάνουμε ότι καταπολεμούμε την φτώχεια και την ανισότητα. Σας παρακαλώ λοιπόν να μου δώσετε μία απάντηση. Σας ευχαριστώ Μπρέσο. Κύριε Πρωθυπουργέ, όπως ε, ήδη κάποιοι συνάδελφοι είπαν και όχι μόνο οι Ιταλοί, εμείς εδώ εργαζόμαστε σε έργα που στόχο έχουν να βοηθήσουν την Ιταλία και την Ευρώπη. Και η γραμμή αυτή, η μεταφορική ε, της Μεσογείου, γιατί δεν είναι μόνο από το Τωρίνο στην Λιόν, είναι αυτή ακριβώς η οποία θα αποκαταστήσει την ισορροπία του συστήματος μεταφορών προς νότον και όταν ολοκληρωθεί θα συνδέσει τα λιμάνια της Μεσογείου και θα επιτρέψει να αναπτυχθούν. Και το είπατε επίσης ε, ότι η κυβέρνησή σας ε, έχει κάνει μία ανάλυση κόστος η οποία όμως δεν λαμβάνει υπόψη το χρονικό πλαίσιο σε βάθος 50 ετών ε, για την απόσβεση. Κύριε ε, Πρωθυπουργέ, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να σκέφτεστε μόνο και σαν Ευρωπαίος και όχι μόνο να σκέφτεστε τα μικρά εσωτερικά ιταλικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ, ε, εγώ θα σας πω ότι είμαι από την Σουηδία, με εκλεγμένη, αλλά είμαι περήφανη που είμαι Ιταλίδα. Αλλά ε, τώρα πια είμαι όλο ένα λιγότερο περήφανη για την Ιταλία μου. Την Ιταλία που εργάζεται, που έχει τεράστια καρδιά, ε, που δεν γυρνάει τις πλάτες όταν τα παιδιά βρίσκονται να κολυμπάνε στη θάλασσα, που κλείνει τα λιμάνια της, που γνωρίζει ότι το κοινό μας μέλλον είναι η Ευρώπη. Εδώ και ένα χρόνο η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος. Την αξιοπιστία τη σε όλα τα μέτωπα. Ανησυχεί η ε, κακοδιαχείριση της οικονομίας που έχει φέρει σε ύφεση την Ιταλία. Οι νέοι, κύριε Πρωθυπουργέ, οι νέοι ζητούν δουλειά. Δεν ζητούν ελεημοσύνη. Θέλουν αξιοπρέπεια και όχι κουβέντε προπαγάνδα. Θέλουν συγκεκριμένε απαντήσει. Τι θα δώσετε συγκεκριμένε απαντήσει, μα ακούτε, ε, στου ανέργου, στην ελάφρυνση του χρέου που οδηγεί στη φτώχεια οικογένεια οικογένειες και επιχειρήσεις. Με ακούτε. Α, ωραία, ευχαριστώ. Ε, και ανησυχεί ακόμα περισσότερο ε, ο εκτροχιασμός προς την εθνική κυριαρχία και τον εθνικισμό της κυβέρνησή σας. Δεν είναι το πρόβλημα η συνεργασία της Ιταλίας με άλλες χώρες. Η Ιταλία είναι μια χώρα σε θέση να χτίζει γέφυρες, όχι να ανοίγει χαντάκια και ε, να προκαλεί ρήξεις. Χρειάζεται αλληλεγγύη, αλλά με διάλογο, όχι με προσβολές. Πα, πα, ε, φτάνει αυτή, αυτό το παράδοξο που λέει ότι οι γειτονέ μα είναι οι πρώτοι μα εχθροί. Δεν θα προχωρήσουμε αν δεν δημιουργούνται ε, συμμαχίε. Ε, δεν θα δημιουργήσουμε σωστά. Μα μας ακούν ο Γκάσπαρη και ο Σπινέλη και μα βλέπουν. Αλλάξτε πορεία, κύριε Κόντε. Σόλτε. Κύριε Σόλτες. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μιλήσω για μια αλληλέγγυα Ευρώπη, μια Ευρώπη της συμφιλίωσης, μια Ευρώπη ενωμένη. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και εσείς ο ίδιος μιλάτε με λόγια που δείχνουν το μίσος σαν τα θύματα να μην ήταν αρκετά στο παρελθόν. Αρνείστε με κάποιο τρόπο την ιστορία. Τα θύματα αυτά έδωσαν τη ζωή τους έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά συμπεριλαμβανομένου και το σύνορο μεταξύ Σλοβενίας και Ιταλίας και πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να παραιτηθείτε μετά από αυτά στα σχόλια. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση. Δυστυχώς Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κυρία Σλάιν, δεν μπορώ να του ικανοποιήσω όλου. Είναι 50 οι βουλευτέ. Έδωσα και παραπάνω χρόνο. Ο καθένα θέλει να μιλήσει. Κύριε Κόντε, παρακαλώ. Απαντήστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ορισμένες παρεμβάσεις έθιξαν θέματα πολιτικού χαρακτήρα. Η πολιτική συζήτηση σκοπό έχει να εξυπηρετεί την ε, δημοκρατική λειτουργία. Ε, ακόμα και αν είναι εντονή, ακόμα και αν κάποιες φορές είναι δυσάρεστες οι αντιπαραθέσεις. Κάποιες παρεμβάσεις δεν θα πρέπει καν να σχολιαστούν, διότι προφανώς νομίζουν ότι θα προσβάλλουν όχι μόνο τον ίδιο τον ομιλόντα αλλά τον ολόκληρο, ολόκληρο το λαό που εκπροσωπεί, που εγώ εκπροσωπώ. Ορισμένοι είχαν το θράσος, και το λέω με απόλυτη επίγνωση, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κάποιοι είπαν και ως επικεφαλής ομάδας, εκπροσωπώντας ολόκληρη πολιτική ομάδα, ότι είμαστε παλιάτσι που εκπροσωπούμε τον Ιταλικό λαό. Εγώ δεν είμαι μαριονέτα, δεν είμαι μαριονέτα ούτε αισθάνομαι έτσι. Είμαι υπερήφανος που εκπροσωπώ έναν ολόκληρο λαό. Είμαι υπερήφανο και καμαρώνω που μπορώ να ερμηνεύσω τη βούληση για αλλαγή των Ιταλών και, των... ολόκληρου του λαού. Είμαι υπερήφανος που μπορώ να συγκεφαλαιώσω την πολιτική γραμμή μιας κυβέρνησης που δεν είναι μαριονέτα, γιατί δεν ακολουθεί λογικές των λόμπι, ούτε επιχειρηματικών κύκλων. Ίσως μαριονέτες είναι αυτοί που ασχολούνται με τα λόμπι, τις επιχειρηματικούς ομίλους και τις τραπεζικές ομάδες μου είπατε ορισμένοι και νομίζω και εδώ ε, ξεφεύγουμε από την έντιμη και έστω και ε, δύσκολη πολιτική συζήτηση ότι υπάρχει ε, και μια κουβέντα που έγινε μεταξύ εμού και της καγκελαρίου Μέρκελ Όποιο ε, τα είπε αυτά μπορεί να ντρέπεται δημοσίως για δικό μου λογαριασμό αν ίσχυαν αυτά τα λόγια. Είπε ότι εκπρόσωπος ενός ε, έχει υψηλά ρεκόρ ε, ως προς την ε, ε, εκτίμηση που του τρέφει το κοινό. Ίσως άλλοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ντρέπονται μεταφέροντας αυτά τα λόγια. Επίσης, και εδώ φτάνουμε στο τρίτο σημείο που κατά την άποψή μα ε, ξεφεύγει από την έντιμη πολιτική συζήτηση, ακόμη και αν αυτή ήταν ε, έντονη, ότι οι υπουργοί μου, υπόθηκε μάλλον, ότι οι υπουργοί μου δεν συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Υπουργικά Συμβούλια. Η κυβέρνησή μου δεν παρίσταται στη συνόδο ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν θα σα θυμίσω τι γίνεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Απλώ να θυμίσω ότι η κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπηθεί και από υφυπουργό, από κάποιον άλλο εκπρόσωπο και ότι ανέκαθεν παριστάμεθα σε όλε τι συνόδου και σε όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια και συμβούλια υπουργών. Το θυμίζω και το τονίζω για να είμαι ακόμη πιο άμεσο και ότι εσείς που εκφράζετε ένα κόμμα το οποίο στο παρελθόν δεν ε, συμμετείχε επαρκώς στην περίπτωση της ΕΜΑ και ακόμα πληρώνουμε τις συνέπειες. Ε, κατά τα άλλα, Πρόεδρε, θα έρθω τώρα στις ερωτήσεις. Vengo και τώρα έρχομαι. Κύριε Ντάντε, σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε λίγο διαφορετική γλώσσα. Ας προσπαθήσουμε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε δύο λεφτά. Παρακαλώ. Πρωθυπουργέ, με συγχωρείτε. Παρακαλώ όλες και όλους μην χρησιμοποιείτε προσβλητικέ εκφράσει. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, μπορείτε να εκθέσετε οποιαδήποτε πολιτική θέση σα αρέσει, αλλά μην προσβάλλετε του άλλου. Και άλλοι εκπροσωπούν ε, ε, το λαό και είναι νομίμω εκλεγμένοι. Μην προσβάλλετε τον Πρωθυπουργό τη Ιταλική Δημοκρατία, ο οποίο έχει προσκληθεί από εμά εδώ. Δεν έχει έρθει ε, με το ζόρι. Τον καλέσαμε. Σας παρακαλώ λοιπόν κόσμια γλώσσα. Απευθύνομαι κυρίω στου συμπατριώτες μου του Ιταλού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ λοιπόν θα έρθω και στα πολιτικά ζητήματα που τέθηκαν, που είναι επίσης πολύ ενδιαφέροντα να απαντήσω σε συγκεκριμένο αίτημα. Μου ρωτήθηκε να πω για την στήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Να θυμίσω στις 29 Ιανουαρίου ήμουν στην Λευκοσία, όπου μαζί με άλλες 7 χώρες της Νοτιού Ευρώπης ε, συζητήσαμε και δώσαμε και μια τελική συνέντευξη τύπου κοινή και είπαμε, τοποθετηθήκαμε συγκεκριμένα. Οπότε υποστήριξη προς την Κύπρο έχει ήδη δοθεί. Σε ό,τι αφορά τα άλλα ερωτήματα, ε, υπόθηκαν πράγματα πραγματικά που προκαλούν ντροπή για την Ιταλία. Ότι αφήνουμε να πεθαίνουν παιδιά στη θάλασσα. Αυτά είναι πραγματικά σοβαρά, είναι ε, απίστευτα αυτά που λέγονται. Το είπα και προηγουμένως έχουμε καθήκον να ενημερωνόμαστε όταν μιλάμε εδώ από αυτά τα έδρανα. Είπα προηγουμένως ότι ανέκαθεν ίσα ίσα που παρενέβημεν για να φροντίσουμε ότι ε, εξασφαλίζουμε την ακαιρεότητα των πιο ευάλωτων ακόμα και σε δύσκολες και πολύ προβεβλημένες υποθέσεις διάσωσης. Κοιτάξαμε πρώτα την ασφάλεια γυναικών και παιδιών, τους μεταφέραμε. Τους ε, αποβιβάσαμε από τα σκάφη, ζωντά τους. Ε, εδώ λοιπόν την αλληλεγγύη τη θεωρούμε κάτι που εκφράζεται στην πράξη. Στην Ευρώπη θα πρέπει να περάσετε από τα λόγια στα, στις, στη δράση. Ε, Όσοι χώρα έχουμε κάνει πολλά. Γαλλία, για το κεφάλαιο Γαλλία. Ε, το είπα επανειλημμένος η Ιταλία είναι υπερήφανη για τον παλιό της δεσμό, οικονομικό και πολιτιστικό κυρίως με τη Γαλλία. Ξεκινά με τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Ποιος το αμφισβητεί. Μιλάτε για διαφωνία, μιλάτε για αντιπαράθεση, για μια συγκεκριμένη υπόθεση και λέτε ότι πάει στην ουσία. Μιλάμε για δύο συστήματα που λειτουργούν παράλληλα και συνδυάζονται, ε, αλληλοδιεκτρέφονται στον, ε, αλληλοτροφοδοτούνται μάλλον στο πολιτιστικό επίπεδο και το οικονομικό. Επίσης, συζήτησα με κάποιους εκπροσώπους του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων Βεβαίως αυτό έγινε στα πλαίσια του ιδιότητα ενός ηγέτη πολιτικής ομάδας. Πρέπει να υπάρχει πολιτική συζήτηση. Πρέπει οι επιλογές να μπορούν να τεκμηριωθούν, ε, οπότε εφόσον τεκμηριώνονται είναι και νόμιμε νόμιμες και θεμητές. Για τη Βενεζουέλα υπόθηκε κάτι που είναι κατάφορα ψεύδος. Ε, η Ιταλία υποστηρίζει το Μαδούρο και η Ιταλία δεν ζητά προεδρικέ εκλογέ. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. δεν υπάρχει, ότι δεν βιαζόμαστε. Οι δηλώσει μου είναι όλε το αντίθετο, λένε. Το καθεστώ του Μαδούρο σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται από την Ιταλία. σα ίσα διακηρύξαμε ε, και αποφανθήκαμε ότι οι προεδρικέ εκλογέ δεν ήταν νόμιμε. Το Ευρωκοινοβούλιο τι αναγνώρισε. Δεν αποστήλαμε τίποτα ε, ω ε, αναγνώριση. Δεν θεωρούμε ότι ο πρόεδρο Μαδούρο έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Ζητάμε όμω το δυνατόν νωρίτερα προεδρικέ εκλογέ. Ελεύθερε. Και το έχουμε πει με κάθε τρόπο εκλογέ ω το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί ο πληθυσμό τη χώρα υποφέρει. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό θα ε, επιτευχθεί εάν ε, υπάρξουν ε, τέτοιε ρήξει στη χώρα και αναγνωριστεί, το είπα, το αξίωμα πρόεδρο κάποιο που δεν έχει κερδίσει νόμιμα εκλογέ. Πρέπει γρήγορα να πάμε σε ταχεία επίλυση του θέματο με δημοκρατικό τρόπο. Επίση, και νομίζω τέθηκε το θέμα της οικονομίας ρωτήθηκε γιατί η Ιταλία δεν δίνει σημασία και στην ευρωπαϊκή διάσταση της βιομηχανικής πολιτικής. Έχουμε αναγνωρίσει τη σημασία του προγράμματος Juncker, το είπα εγώ ίδιος. Ανέκαθεν υποστηρίζαμε την σημασία και την αξία μιας βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρώπη, από την Ευρώπη. Ε, μάλιστα, έχουμε υπογραμμίσει την σημασία ενός προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Ε, προπολογισμού που θα έχει και μια λειτουργία σταθεροποίησης. Και για να παραμείνουμε στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής και της κοινωνικής πολιτικής, η χώρα μας, κοιτάξτε, είπατε, δεν αναπτύσσεστε. Τι θα πει αναπτυσσόμαστε. Θα πρέπει να βασιστούμε σε πολιτικούς υπολογισμού του παρελθόντος. Μήπως είναι ακόμα λίγο νωρί. Μήπως είναι ακόμα λίγο νωρί για να αξιολογήσουμε ο οικονομικός ελιγμός που κάνουμε τώρα, η αλλαγή πορείας που ακόμα πραγματοποιείται, θα δώσει καρπούς. Εγώ έχω αναπτύξει ένα σκεπτικό ότι η οικονομική ανάπτυξη θα γίνει στο δεύτερο εξάμεινο, θα φαίνεται στο δεύτερο εξάμεινο το 2019, διότι ακριβώς και πολύ απλά η οικονομική μας πολιτική, τα μέτρα μας δεν μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως αυτούς τους πρώτους μήνες του έτους. Ε, να έχετε υπόψη ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά το σύστημα παραγωγής. Πώς θα μπορούσαμε να μην ασχολούμαστε με το πρόγραμμα επενδύσεων το είπα και προηγουμένως. Και κάποιοι είπαν κάτι εντελώ λανθασμένο. Βεβαίω και εργαζόμαστε από αυτού. Και χθε μόλι, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, εγώ ο ίδιο βρισκόμουν στην περιοχή τη Νότια Ιταλία, την περιφέρεια αυτή, όπου είναι μεγαλύτερη οικονομική ύφεση σε σχέση με αλλού, και για σκοπού κοινωνική ανάπτυξη υπέγραψα τρει ε, συμβάσεις στο Μολύζε, τη Σαρδινία και την Παζιλικάτα για σκοπούς κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό έχει πραγματιστικό σκοπό. Θέλουμε να στηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη με όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Ακόμη και το εισόδημα, το ελάχιστο εισόδημα για τους πολίτες, για τους φτωχότερους πολίτες. Θα μπορούσε να είναι σοσιαλιστικό τέχνασμα. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Όλοι το συζητάνε αυτό το μέτρο γιατί έχει καταλητικό χαρακτήρα για τις δημόσιες συζητήσεις. Εδώ όμω είναι υπαρξιακό το θέμα, διότι είναι και θέμα προπολογισμού και κυρίως το συλλάβαμε στο επίπεδο ενός συμφώνου εργασίας, κοινωνικής συμπερίληψης, για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε στο χώρο της, αγο... της εργασίας και της παραγωγής 5 εκατομμύρια φτωχούς. 5 εκατομμύρια φτωχούς ε, στους οποίους απευθύνεται απευθείας αυτό το μέτρο είναι εντελώ εκτό συστήματο, οποιοδήποτε κοινωνικού παραγωγικού μηχανισμού, εκτό του χώρου τη εργασία. Χωρί το άρθρο 3, στο δεύτερο εδάφιο του υπέροχου συντάγματό μα, του συντάγματο τη Ιταλία, δεν θα έχουν καμία ε, ηλική, καμία χειροπιαστή πραγματικότητα να συμμετέχουν στην ε, δημοκρατική, κοινωνική και πολιτική ε, διαδικασία και το γίγνεσθε τη χώρα μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ εγώ κύριε Πρωθυπουργέ, εκπρόσωπε του, της Ιταλικής κυβέρνησης, της ε, Δημοκρατίας της Ιταλίας. Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας και τις απαντήσεις σας. Με συγχωρείτε κάποιες φορές το ύφος που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν κατάλληλο, αλλά στην Ολομέλεια πάντοτε είναι έντονες οι συζητήσεις, γεμάτες πάθη, όταν υπάρχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα τα οποία συζητούμε. Πάνω από όλα σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ένωσής μας.